So, liebe Kolleginnen, Kollegen und meine Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, παρακαλώ καθίστε, έχουμε ήδη καθυστερήσει λίγο. Σας ε, καλωσορίζω όλους ε, στην ακρόαση για την ε, μεταρρύθμιση της διπλής χρήση. Είμαι σίγουρος ότι με το θέμα αυτό ασχολούμαστε με ένα θέμα σημαντικό και ευαίσθητο ζήτημα της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας το οποίο αφορά την ε, συνέχεια, την συνέπεια και την διαφάνεια και έχουμε κάνει μια κοινή δήλωση Συμβουλίου, Κοινοβουλίου και Κομισιών γιατί ζητήσαμε μια επαναπροσέγγιση του θέματος και η Κομισιόν 28 Σεπτεμβρίου κατάσε μια νομοθετική πρόταση που προβλέπει κάποιες ε, ουσιαστικές αλλαγές σε σχέση με την προηγούμενη, ειδικά όσον αφορά τα κριτήρια τήρησης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και όσον αφορά τους μηχανισμούς ελέγχου και την εναρμόνιση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, δεν θα πω τίποτα άλλο για να έχουμε αρκετό χρόνο να ακούσουμε τους ειδικού. Που είναι άλλωστε το βασικό θέμα της ακρόασης. Για να δούμε ακριβώς ε, τι μπορούν να μας πούν. Έχουμε χωρίσει αυτή την ακρόαση σε δύο μέρη. Πρώτον, για να σκεφτούμε ποιες προκλήσεις ε, και απειλές ε, έχουμε με το θέμα της διπλής χρήσης ε, και των εξαγωγικών περιορισμών, ειδικά από πλευράς πληροφόρησης και επικοινωνίας και δεύτερον, συγκεκριμένα να συζητήσουμε πώς θα μπορέσουμε να διαμορφώσουμε αποτελεσματικότερη την νομοθεσία. Στο πρώτο πάνελ χαίρομαι που έχουμε μαζί μας τον κύριο Μπεν Βάγνερ του Ινστιτούτου Επιστήμης και Πολιτικής ε, από τη Γερμανία, την κυρία Λουσί Κραχούλτσοβα από το Access Now και τον κύριο Μάγνους Νορντέους από την Έριξον. Ακριβώ ειδικού δηλαδή ε, πάνω στα θέματα αυτά της τηλεπικοινωνίας και των υπολογιστών. Ο καθένας λοιπόν έχει 7 λεπτά χρόνο και ξέρετε πως ε, τα τηρώ εγώ αυτά. Λοιπόν, θα δώσω πρώτα απ' όλα τον λόγο στον κύριο Βάγνερ. Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ και για την πρόσκληση που μου απευθύνατε. Είμαι από το Γερμανικό Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων και να κάνω κάποιες παρατηρήσεις από την δική μου την προσωπική σκοπιά για το ότι θεωρούμε εμείς ότι είναι τα βασικά ζητήματα της ε, διπλής χρήσης. Λοιπόν, γιατί βρισκόμαστε εδώ. Ο λόγος για τον οποίο είμαστε εδώ σήμερα, αν δεν βλέπετε τις διαφάνειες έχετε μία ιδέα, είναι το ότι παρόλες τις συζητήσεις για το θέμα έχουμε μια κατάσταση όπου εξάγονται τεχνολογίες ε, επιτήρησης από ευρωπαϊκές χώρες εδώ και πολλά χρόνια και παρά τις προσπάθειες εξακολουθεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Δεν ήμασταν σε θέση να μειώσουμε αυτή την διάδοση μέσω κανονισμών ελέγχου των εξαγών και παρά τα όσα γράφουν διάφοροι δημοσιογράφοι, κυρίως στην Ευρώπη, βλέπουμε πως ακόμα και όταν καλύπτονται από εξαγωγικούς ελέγχους, η αποτελεσματικότητα αυτών των ελέγχων είναι περιορισμένη. Έχουμε λοιπόν μια κατάσταση όπου το υφιστάμενο ρυθμιστικό πλαίσιο δεν είναι τελείο και έχουμε ανησυχίες. Και αυτό το οποίο προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για όσους δεν το γνωρίζουν, ουσιαστικά βασίζεται στην έννοια της ανθρώπινης ασφάλειας που αφορά διάφορα θέματα στην ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική και η προσέγγιση αυτή η ίδια νομίζω δεν είναι κάτι το επίμαχο. Έχει ενσωματωθεί σε πολλές πτυχές του ΟΗΕ, είναι κάτι το φυσιολογικό. Είναι ένας υφιστάμενος μηχανισμός βεβαίως. Το θέμα δεν είναι το εάν αλλά το πώς. Και αυτό ακριβώς θα συζητήσουμε τις ώρες που έρχονται ειδικά όταν περνάμε από πτυχές όπως η προσέγγιση ανθρώπινης ασφαλείας ε, στις ε, ληφθείς του ΟΗΕ. Λοιπόν, από τη δικιά μας σκοπιά μας στιγμής έχουμε την συνεννόηση Βασενάρ που είναι ο βασικός μηχανισμός σε διεθνές επίπεδο έτσι ώστε να υπάρχει κάποιο συντονισμός για τα είδη διπλής χρήσης. Και όπως ξέρετε ε, δεν είναι κάτι το δεσμευτικό. Τι σημαίνει αυτό λοιπόν, ότι τα κράτη-μέλη της Ένωσης αποφάσισαν να κινηθούν μόνα του όταν θέλουν να καινοτομήσουν για τα είδη διπλού ελέγχου. Δηλαδή η Γαλλία και η Γερμανία ανέπτυξαν κάποιες αλλαγές ε, από μόνος τους, ε, άρα υπάρχει ένας μηχανισμός ο οποίος δεν είναι η βάση, αλλά δεν είναι και μηχανισμός στο εθνικό επίπεδο. Και νομίζω ότι παρέχει έτσι μια ευκαιρία να υπάρξει ένα περαιτέρω επίπεδο πολυμερών συμφωνιών έτσι ώστε τα κράτη-μέλη και οι ανησυχίες που έχουν ε, να μπορούν να ελεγχθούν σε πολυμερές και όχι απλά επίπεδο. Τώρα, για να περάσουμε στην ίδια την πρόταση, υπήρχαν κάποιες ανησυχίες ε, για το θέμα αυτό και για το θέμα της διπλής επιμέλειας και το ότι οι εταιρείε αν είχαν συγκεκριμένη γνώση παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα έπρεπε να ζητήσουν κάποια άδεια. Και νομίζω ότι εκεί το ζήτημα είναι ότι πρέπει να γνωρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη έχει αναλάβει δεσμεύσει ε, για επιχειρήσεις ε, οι οποίες θα αναλάβουν ε, την επιμέλεια αυτή. Είναι κάτι το σύνηθες που κάνουν οι εξαγωγείς. Δηλαδή πρέπει να συμμορφώνουν ο πελάτες τους σε πολλά και διάφορα πράγματα και βεβαίως το θέμα είναι σε ποιο βαθμό θα προχωρήσουμε, αλλά το γεγονός πως η δέουσα επιμέλεια είναι κάτι το ασύνηθες, νομίζω δεν ισχύει ταυτόχρονα. Για να προχωρήσουμε αυτά τα οποία έχουν συζητηθεί εδώ πέρα, να βλέπουμε την ίδια πρόκληση, το ίδιο θέμα, εάν οι εταιρείε έχουν κάποιες θετικές ε, γνώσεις, ε, τότε ότι δηλαδή θα υπάρξει τέτοια χρήση για παραβιάση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τότε πρέπει να ζητήσουμε μια άδεια και ενώ και πάλι μπορούμε να ζητήσουμε ακριβώς, να, συζητήσουμε την διατύπωση, νομίζω ότι η αρχή είναι σαφής. Εάν δει κάποιο ότι οι τεχνολογίες του μπορεί να χρησιμοποιηθούν με τρόπο που δεν θα έπρεπε, θα πρέπει να φροντίσει να κινείται εντός του νόμου. Βεβαίω αυτό δεν ισχύει για τεχνολογίες ε, που αφορούν ε, την έρευνα, αλλά νομίζω ότι το σκεπτικό είναι λογικό και δεδομένου του ότι έχουμε κάποιες γενικές εφαρμογές σε ευρωπαϊκό επίπεδο, παραδείγματος χάρη όταν μιλάμε για όπλα μαζικής καταστροφής, υπάρχει το ερώτημα το αν μπορούν να εφαρμοστούν για αυτούς τους τομείς, πώς μπορούμε να πούμε, πώς μπορούμε να πούμε ότι για άλλους τομείς είναι αδύνατον. Δεν νομίζω. Όμως, αν είναι να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής, πρέπει επίσης να αναγνωρίσουμε ότι έτσι δημιουργείται ένα έλλειμμα λογοδοσίας. Δηλαδή, αν δίνουμε μεγαλύτερη διακριτική ευχέρεια στις εφαρμοστικές αρχές, ε, πρέπει να διασφαλίσουμε και μεγαλύτερα επίπεδα λογοδοσίας. Είναι μια κλασική κατάσταση όπου αυξάνει τη διακριτική ευχέρεια των θεσμικών οργάνων, οπότε πρέπει να αυξηθεί και η λογοδοσία. Και αυτό βεβαίως δεν σημαίνει μόνο λογοδοσία, αλλά και διαφάνεια. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή πολλές διαφορετικές εφαρμογές σε επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου διαφορετικά κράτη-μέλη έχουν διαφορετικά επίπεδα διαφάνειας και υπάρχει ανάγκη διαφάνεια για ίσους όρους ανταγωνισμού, αλλά και για να διασφαλίσουμε ότι, και όπου βρισκόμαστε τώρα, γνωρίζει το κοινό τι αποφάσεις λαμβάνονται και είναι σε θέση να συμφωνήσει, να διαφωνήσει. αν δεν θα πρέπει να πάμε σε μια κατάσταση όπου θα είναι σαφές το ποιες είναι οι αποφάσεις και έρχομαι έτσι στις τελευταίες διαφάνειες για να έχετε μία ιδέα. Το θέμα δεν αφορά μόνο την διαφάνεια, αφορά και την κρυπτογράφηση. Όταν μιλάμε για κλάδους που πρέπει να προστατεύονται, πρέπει να διασφαλίσουμε στο πλαίσιο των συζητήσεων που έχουμε ότι δεν θα βλάπτουμε την έρευνα ασφαλείας, πράγματα τα οποία θα κάνουν το διαδίκτυο πιο ασφαλές, αλλά και συγκεκριμένες τεχνολογίες όπως η κρυπτογράφηση που είναι από τα πράγματα τα οποία μας επιτρέπουν να συνεργαζόμαστε και να έχουμε ψηφιακές επικοινωνίες πρέπει να είναι ασφαλής και βέβαια κάτι το οποίο είναι σημαντικό για τα μέλη της Επιτροπής σας η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει προδιαγραφές ειδικά για το διεθνές εμπόριο και μην ξεχνάμε πως ε, όταν υπάρχουν διαμαρτυρίες για το παγκόσμιο εμπόριο υπάρχουν γιατί ο κόσμος δεν πιστεύει στις αξίες, ότι υπάρχουν αξίες πίσω από αυτό. Γι' αυτό τώρα είναι μια ευκαιρία για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δείξει ότι στηρίζει τις αξίες στο διεθνές εμπόριο. Και αν υπάρχει διεθνές εμπόριο θα πρέπει να γίνεται με τον σωστό τρόπο. Αυτά και σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Σας ευχαριστώ η κυρία Καχούλκοβα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καχούλτσοβα, είμαι Τσέχα. Σας ευχαριστώ για τα ωραία σας λόγια. Νομίζω ότι ο προηγούμενος ομιλητής έθεσε τα βασικά ζητήματα που θα θέταμε και εμείς ως εκπρόσωποι της, μη κυβερ... Ε, ως εκπρόσωποι της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών. Το ερώτημα που τίθεται είναι πώς θα ε, ε, θωρακίσουμε τους κανονισμούς για τις εξαγωγές και πώς θα ε, συνεχίσουν να λειτουργούν αποτελεσματικά και σε βάθος χρόνου. Τρία μηνύματα θέλω να σας στείλω σήμερα. Πρώτον, χρειαζόμαστε ισχυρή αξιολόγηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεύτερον, να εδραιώσουμε τη διαφάνεια και τις δυνατότητες εντοπισμού των λαθών και παραβάσεων και παρατυπιών. Τώρα, τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να συνάδουν με κριτήρια αξιολόγησης, να είναι συνδεδεμένα. Έχουμε πάρα πολλή νομολογία από το δικαστήριο. Έχουμε την υπόθεση Ζαχάροφ, την απόφαση τέλετου. Να δούμε πώς όλες αυτές τις νομολογίες και τις αποφάσεις θα τις μετεουσιώσουμε σε ε, έννοιες που θα διέπουν τον τρόπο με τον οποίο η ψηφιακή τεχνολογία επηρεάζει τη ζωή μας. Επανειλημμένως ακούμε και λέμε ότι δεν υπάρχει ανάγκη να περιορίσει κανείς ή να ελέγξει την εξαγωγή τεχνολογίων ε, μεταξύ ρυθμιστικών αρχών στην Ευρώπη και αυτό είναι κάτι που μας ανησυχεί. Γιατί πάρα πολλή τεχνολογία ήδη ε, δοκιμάζεται σε εθνικό επίπεδο και εμεί ω Access Now, ω ε, διεθνή παγκόσμια οργάνωση, το βλέπουμε αυτό. Καλό είναι να έχουμε ψηλά στάνταρ για το μήνυμα που στέλνουμε και στου εξωτερικού παρατηρητέ. Έτσι όπως έχει ο κανονισμός δεν είναι σαφές με ποιες συνθήκες ο κίνδυνος για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι αρκετά σοβαρός για να οδηγήσει σε ανάκληση της άδειας. Λέμε serious, λέμε extreme, ε, ε, σοβαρές, ακραίες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ανθρώπινα παραβιώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων πολύ απλά. Δεν μπορούμε να αντικαθιστούμε τον έναν όρο με έναν άλλον όρο. Οι καθοδηγητικές αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, έχουν πολύ σωστή διατύπωση και θα πρέπει να τη συμπεριλάβουμε. Είναι κάτι που για το οποίο ευθύνεται ο ΙΕ και όλα τα μέλη του. Άρα και εμείς προσυπογράφουμε και μπορούμε να το εγγράφουμε. Και έχουμε και ένα έγγραφο το οποίο θα κυκλοφορήσουμε που θα περιλαμβάνει τις πηγές για λόγους βιβλιογραφικούς. Τα κριτήρια αξιολόγησης πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους το, το, τις επιδόσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα του τελικού χρήστη της τεχνολογίας. Ε, και δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο που θα ρυθμίζει τη χρήση της τεχνολογίας από τον τελικό χρήστη. Έχουμε τη διάταξη Access to Remedy στα Ηνωμένα Έθνη, πρόσβαση στα επανορθωτικό μέσα και πρέπει να το περιβάλλουμε, να το περιλάβουμε εδώ. Υπάρχει απειλή για την ανθρώπινη ασφάλεια αλλά και για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ποιο νομικό πλαίσιο έχουν οι άνθρωποι στην εκάστοτε χώρα όπου θα χρησιμοποιηθεί αυτή η τεχνολογία για να τους προστατεύσει. Πολύ συχνά στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε ένα χι πλαίσιο και μετά εξάγουμε το ένα κείμενο και τελικά δεν ε, υπόκειται ο λαός της τρίτης χώρας όπου εξάγαμε τεχνολογία στα ίδια επανορθωτικά μέσα και στις ίδιες δυνατότητες εάν πληγούν τα δικαιώματά του. Άρα θέλουμε πιο ισχυρό ε, κείμενο και μια τεχνολογία catch all. Να βελτιώσουμε τη τεχνολογία εποπτείας, επιτήρησης, παρακολούθησης, ενδεχομένως όλα αυτά είναι προβληματικά. Το catch all ε, είναι μια ευκαιρία να είμαστε πρωτοπόροι, να θέσουμε εμείς τα πρότυπα. Όμως, επαφίεται στη διακριτική ευχαίρεια του καθενός να καταγγείλει σοβαρές καταστρατηγίες ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κατά πόσο η τεχνολογία χρησιμοποιήθηκε επί σκοπού, με σκοπό να καταστρατηγηθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα ή απλά η τεχνολογία διευκόλυνε στην καταστρατήγηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρέπει όλα αυτά να τα διευκρινίσουμε για να μπορούμε να πάμε σε εταιρείε και να πούμε εδώ παραφερθήκατε και βγήκατε εκτός γραμμής. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά και είναι καλό να γίνεται διαβούλευση με την οργανωμένη κοινωνία των πολιτών, με τον πανεπιστημιακό κόσμο, με όσους ενδιαφέρονται. Σε κάθε περίπτωση έχουμε πάρα πολλούς υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων που ε, δημιουργούν υλικό νομικό, Privacy International, Citizen Lab, το εργαστήριο των, ε, ε, των πολιτών, το να το αγνοεί κανείς είναι κρίμα, γιατί είναι δύσκολο να το βρούμε, να το ότι υπάρχουν πληροφορίες και έχει γίνει πολύ σοβαρή δουλειά από τις οργανώσεις επιτόπου και τους ε, ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων επιτόπου μπορούμε να βασιστούμε στη βιομηχανία ότι θα αυτορυθμιστεί, εγώ είμαι κατά. Είναι πολύ μεγάλη ανάγκη για την ευθύνη για τη δέουσα επιμέλεια και οι, αρχές που δίνουν την άδεια θα πρέπει να μπορούν να ελέγχουν την αξιολόγηση που η ίδια η βιομηχανία κάνει για τον εαυτό τους και γι' αυτό έχουμε το catch all η τρομοκρατία ορίζεται πολύ διαφορετικά από τη μία χώρα στην άλλη. Η συμπερίληψη της τρομοκρατίας σε αυτόν τον κανονισμό είναι ε, πολύ δυστυχής και θέλουμε να διαγραφεί από το catch-all regulation. Και τέλος, ένα από τα βασικά που μπορούμε να κάνουμε με αυτή την αναθεώρηση είναι η διαφάνεια, η λογοδοσία να συνδεθούν άρεκτα με τη διαδικασία ελέγχου των εξαγωγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο συνασπισμός, η συμμαχία εναντίον της ε, μη νόμιμης εποπτείας των εξαγωγών έχει καταλήξει σε ένα έγγραφο και ε, αναφέρεται σε ευρήματα και πολύ σημαντικά. Στο κείμενο υπάρχει μια διάταξη να υπάρχει αιτήσια αναθεώρηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Νομίζω ότι μέρο τη αναθεώρηση θα πρέπει να είναι ένα φόρουμ και να προσκληθούν εκεί οι οργανώσει ε, τη κοινωνία των πολιτών για να παρουσιάσουν στοιχεία, να ακουστεί η φωνή τους. Ε, Εμεί δεν έχουμε φωνή, δεν ακούγεται και είναι πολύ σημαντικό να αποκτήσουμε. Και κάτι που θα πρέπει να προκύψει είναι η δημοσίευση των στατιστικών για τις συναλλαγές και για τις αιτήσει που ε, υποβάλλονται. Θα σας δώσω το προσχέδιο των βιβλιογραφικών παραπομπών. Βλέπω ότι με διακόπτωται λόγω έλλειψης χρόνου. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα ο κύριος Μάγνους Νορτέος από την Ericsson και Digital Europe. Thank you, So, thank you. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριοι βουλευτές και στο υπόλοιπο ακροατήριο που με ξανακαλέσατε. Την ε, περασμένη φορά, το 2015, είχα πάλι τον ίδιο προγνώμονα δίπλα μου. Εργάζομαι στην Ericsson και είμαι και διευθυντής του, της ομάδας Digital Europe. Ε, προσωπούμε τις εταιρείες IT, ICT της Ευρώπης. Η δική μας άποψη όπως όλοι οι υπόλοιποι πιστεύουμε ότι αυτός ο κανονισμός θα ανοίξει το δρόμο, θα ε, στρώσει το δρόμο για τα επόμενα δέκα χρόνια και τις εξαγωγές της Ένωσης. Πρόκειται για ένα περιβάλλον πολύ περίπλοκο, με ε, λεπτομέρειες τεχνικές με την ε, διάδραση και τις διασυνδέσεις μεταξύ ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής, θα κάνω λοιπόν ό,τι καλύτερο μπορώ για να δώσω μια επισκόπηση της δικής μας της προοπτικής και των προτεραιοτήτων μας. Πρώτα απ' όλα, μετά την ε, επίτευξη της συμφωνίας ITA πέρσι, Είχαμε μια από τις μεγαλύτερες συμφωνίες παγκοσμίως με 80 χώρες ε, να συμφωνούν στη μείωση των δασμών για τα προϊόντα ICT Και αυτό λόγω των θετικών επιδράσεων της χρήσης των προϊόντων αυτών. Ε, γι' αυτό λήφθη αυτή η απόφαση και είναι και κάτι το πρωτοφανές. Σήμερα μιλάμε για την ίδια κατηγορία προϊόντων, αλλά πάλι προπτική. Τώρα σκεφτόμαστε πώς να ελέγξουμε και να περιορίσουμε τη διακίνηση αυτών των προϊόντων. Όμως μην ξεχνάμε τον καθοριστικό όλο της ψηφιακής μηχανίας όταν μιλούμε για αυτά τα προϊόντα. Απευθύνω έκκληση λοιπόν προς όλους τους ενδιαφερομένους να κοιτάξουν ο έλεγχος να μην είναι υπερβολικός ώστε να επιτρέπεται η διαχτή σύνδεση μέσω του διαδικτύου των πραγμάτων και να χρησιμοποιηθούν οι ρηξικέλευτες ε, τεχνολογικές λύσεις που επιτρέπουν να γίνει τεράστια πρόοδος σε όλες τις χώρες. Δεν πρέπει εξαγωγές να απορρίπτονται, εκτός αν υπάρχουν βάσιμοι πολύ σοβαροί λόγοι. Κατά την άποψή μας, καμία χώρα δεν μπορεί να παρακάμψει τους ελέγχους και θα πρέπει να δούμε τις επικρίσεις μας προς τους Αμερικανούς νομοθέτες που επιβάλλουν πολλές φορές υπερβολικά πολλούς ελέγχους και περιορισμούς, να μην κάνουμε τα χειρότερα. Οι τεχνολογικές εξελίξεις συνεχίζονται. Πρέπει λοιπόν στις εξαγωγές να δώσουμε νομική ε, βεβαιότητα με σαφέστατους ορισμούς με τους οποίους όλοι να συμφωνούμε από ό,τι άκουσα και από τις άλλες παρουσιάσεις. Στην ε, συζήτηση που γίνεται φέτος ακούσαμε ότι η έλλειψη σαφήνειας και νομικής βεβαιότητας είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της βιομηχανίας. Αλλά το εντόπισαν όλοι οι ενδιαφερομένοι, όχι μόνο εκπρόσωποι των εταιριών. Πριν ε, περάσουμε σε σαφέστερους ορισμούς, να ε, ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που αναγνωρίζει το σοβαρό ρόλο της κρυπτογράφησης των ε, κάποιων δεδομένων. Η κρυπτογράφηση είναι ε, ένα από τα σοβαρότερα μυστικά, αλλά σε αυτό θα πρέπει να έχει πρόσβαση ο καθένα. Η βουλευτή σα εδώ, η κυρία Σχάκε, είπε ότι θα πρέπει να υπάρχει στον κατάλογο περιγνωμόνων δυνατότητα να καθορίζεται ποιο θα έχει δικαίωμα κρυπτογράφηση. Η δική μου απάντηση είναι όχι για την κρυπτογράφηση θα πρέπει να κοιτάξουμε να μην έχουμε τόσου περιορισμού για να υπάρχει λιγότερο διοικητικό άχθο για τι εταιρείε και να είμαστε όλοι στο ίδιο επίπεδο για την ε, διαχείριση των ίδιων προϊόντων. Επίσης, η μεταφορά της τεχνολογίας και του λογισμικού εντός ενός συγκεκριμένου ομίλου ε, θα πρέπει να γίνεται με μια ειδική διαδικασία διοδότησης που και αυτή εκτιμάται ιδιαίτερως. Τώρα η αρχική μου ανησυχία διαβάζοντας την πρόταση της Επιτροπής επιβεβαιώνεται κάπως από τη μελέτη αντικτύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που λέει ότι εξ exposed έλεγχη και ενδεχόμενες τρευλώσεις του ανταγωνισμού θα αντιμετωπίζονται στο κατάλληλο επίπεδο. Τα θέματα αυτά όμως ούτως ή άλλως επιλύονται σε διεθνές επίπεδο. Οπότε οι έλεγχοι θα πρέπει να γίνονται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο στο διεθνές επίπεδο. Για να είναι αποτελεσματικά όλα αυτά και να μην υπάρχει στρέβλο στον ανταγωνισμό, οι ε, ε ελεγκτέ των εξαγωγών τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να βασίζονται στι δεσμεύσει και τι ε, ε, υποχρεώσει των κρατών μελών. Και ο νέο ορισμός της διπλής χρήση το άρθρο 2 ε, με την ε, παράμετρο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δίνει μια νέα διάσταση. Η κοινότητα ελέγχου των εξαγωγών έχει αλλάξει αρκετά και λαμβάνει υπόψη τον ορισμό της διπλής ε, χρήσης. Πρόσφατα είχαμε έναν Ιάπωνα εμπειρογνώμα από το θέμα εδώ στις Βρυξέλλες και είπε ότι θέλει να υπάρξει αυτή γράμμιση με τον ε, κατάλογο ελέγχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να ωφεληθούν και οι εταιρείε και όλη η κοινότητα των ελεγκτών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως δεν είναι πάντοτε αντιληπτή, δεν γίνεται πάντοτε αντιληπτή ως υπόδειγμα. Έχουμε ένα παράδειγμα από τη Σιγκαπούρη, όπου έπαψε να εφαρμόζει το κατάλογο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, διότι δεν ε, λειτουργούσε πλέον ε, αποτελεσματικά, οπότε θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει υπόψη και τις διεθνείς διαστάσεις του θέματος. Επίση, θα πρέπει η δέουσα επιμέλεια με σχετικά προγράμματα να ενισχυθεί το ίδιο και σχετικά προγράμματα στι επιχειρήσει για να λαμβάνουν υπόψη και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Στι όλε μα προσπάθειες περί ηθικής ε, θέσαμε τα θέματα αυτά, αλλά αν η διπλή χρήση προχωρήσει και μιλάμε και για ανθρώπινα δικαιώματα, είναι σημαντικό να ξέρουμε πού στοχεύουμε και πού όχι, σε ποιου, δηλαδή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ε, δημοσίευσε ένα κατάλογο με τους προβλεπόμενους τελικούς χρήστες και σε συνεργασία με τους άλλους φορείς όπως την ESIA ε που θα πρέπει να δώσει παραδείγματα από συγκεκριμένα κράτη-μέλη και το τι συμβαίνει εκεί για να αιτιολογηθούν οι προτάσεις. Τα διαφορετικά συστήματα κυρώσεων, οι νομοθεσίες περί καταδίκης των βασανιστήριων, όλα αυτά θα πρέπει να προχωρήσουν, αλλά να υπάρχει και συνδυασμό με τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Ο εξαγωγέας θα έχει την υποχρέωση να ορίσει ο ίδιος και να εντοπίσει ο ίδιο τον τελικό χρήση, ενώ νομικό δεν είναι υπεύθυνο για κάτι τέτοιο. Βλέπω ότι ο χρόνο μου τελειώνει, οπότε θα ολοκληρώσω. Το συμπέρασμα μας είναι ότι το εξαγωγικό μας σύστημα θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί με άλλα εξαγωγικά συστήματα που ισχύουν και η πρόσβαση στην αγορά ε, είναι ένα κίνητρο, μια ε, κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη. Θα πρέπει λοιπόν να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία της διπλής χρήσης για τις εξαγωγές, αλλά να, σαφή, να βεβαιωθούμε ότι θα παράσχεται η απαραίτητη νομική βεβαιότητα μέσω των σαφέστατων ορισμών, όπω τον παραβιάζει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη δέουσα επιμέλεια και ούτω καθεξή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τώρα θα παρακαλέσω τους βουλευτές να κάνουν ερωτήσεις. Γιατί δεν έχει νόημα να κάνετε δηλώσεις, αλλά να κάνουμε ερωτήσεις στους ειδικού μας. Και ίσως μπορείτε να μας πείτε και σε ποιον ειδικό θέλετε να κάνετε ερώτηση. Πρώτα απ' όλα θα κάνω ερώτηση, θα ζητήσω με συγχωρείτε, από τον συγκριτή και τους κοιόδες συγκητές αν έχουν ερωτήσεις. Κύριος Μπούχνερ, έχετε ερωτήσεις για τους ειδικού, παρακαλώ. Ακριβείς και συγκεκριμένες. Ευχαριστώ. Η πρώτη μου ερώτηση απευθύνεται στον κύριο Βάγνερ. πώς ε, μπορούμε ε, να το πραγματοποιήσουμε, Μιλήσετε για μια ρήτρα catch all. Πώς το βλέπετε σε σχέση με την ασφάλεια προγραμματισμού των επιχειρήσεων. Το δεύτερο ερώτημα αφορά την κυρία Καρχολτσόβα. πώς θα συμπεριλάβετε την κοινωνία των ε, πολιτών. Ότι θα πρέπει να λάβουν μέρος είναι σαφές, αλλά δεν είναι σαφές για μένα η διαδικασία. Πώς ε, μπορούμε να την επισημοποιήσουμε. Και τέλος, για τον κύριο Νορντέους, δεν έχω καταλάβει, ε, απαιτείται έναν πιο ακριβή ε, ορισμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την δέουσα επιμέλεια κτλ. Είναι σαφές ότι πρέπει να ξεκαθαρίσει, αλλά ε, το απαιτείται και για έναν πιο ακριβή ορισμό των αγαθών. Και αυτό είναι πρόβλημα για μένα, γιατί ε, η τεχνολογία αναπτύσσεται πάρα πολύ γρήγορα. Ίσως μπορούμε εντό κάποιου πλαισίου να μιλήσουμε για κατηγορίες, αλλά και αυτό... Ε, εξαρτάται, γιατί βεβαίω η εξέλιξη φεύγει και εκτό των κατηγοριών. Υπάρχουν νέε κατηγορίες. Τι θέλετε ακριβώ να κάνουμε. Ευχαριστώ Φιέλνερ για το ΕΛΚ. Ευχαριστώ. Έχω πολύ συγκεκριμένες ερωτήσεις. Μία για τον κάθε πανελίστα. Πρώτα απ' όλα για την δέουσα επιμέλεια. Ε, ήδη δύο φορές έχω εμπλακεί σε σχετική νομοθεσία για την λάθρο υλοτομία και για τα ορυκτά. Και βεβαίω όλοι θέλουμε σαφήνεια στους νομικούς ορισμούς, ειδικά όταν μιλάμε για κυρώσεις. Οπότε, εντάξει, μιλάμε πολύ καιρό για τον ορισμό της παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τώρα ακούω ότι θα πρέπει να τα αλλάξουμε λίγο ε, και να μιλήσουμε για διευκόλυνση παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μπορείτε λοιπόν έτσι αυθορμήτως να μου δώσετε τρία παραδείγματα προϊόντων πληροφορικής που δεν θα μπορούσαν να διευκολύνουν παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρώτη ερώτηση. Και κάτι άλλο για το catch all. Εντάξει, αντιλαμβάνομαι το, ότι είναι ασαφής ο ορισμός της τρομοκρατίας και το αντιλαμβάνεται ο καθένας διαφορετικά. Τι θα λέγατε για την διευκόλυνση παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν ξέρω. Ισχύει και εκεί κάτι τέτοιο. Δεύτερον, κάτι άλλο το οποίο θα ήθελα να ρωτήσω. Στον κύριο Βάγνερ υπάρχουν παραδείγματα του Κέτσολ πέρα από την ε, κυβερνοπαρακολούθηση γιατί όταν το έλεγξα η αξιολόγηση αντικτύπου της Κομισιόν ε, μόνο για αυτή την αναγκαιότητα μιλούσε. Και βεβαίω έτσι όλοι μιλάμε για κλάδους όπου έχουμε πολύ μεγάλη μεταφορά τεχνολογίας, αλλά προτείνεται τώρα εδώ να ισχύσει στα πάντα. Μπορείτε να μου εξηγήσετε γιατί θα ήταν αναγκαίο πέρα από τον τομέα της ε, κυβερνοεπιτήρησης. Και τέλος, στον κύριο Νορντέους. Μιλάμε επίσης για κάποια αυτόνομη λίστα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά κάποιες φορές έχουν πάει πέρα από την υφιστάμενη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Πώς έχει επηρεάσει αυτό τον κλάδο, ποιος είναι ο αντίκτυπος ε, στην, στην πράξη, το ότι κάποιες χώρες προχώρησαν ε, παραπέρα, έχει υπάρξει κάποιος αντίκτυπος και ποιο θεωρείτε ότι θα είναι ο συνολικό αντίκτυπο του να πάμε πέρα από το εφιστάμενα καθεστώτα. Σας ευχαριστώ. Μπέρντ Λάγκε για τους σοσιαλδημοκράτες, εγώ δηλαδή, για τον κύριο Βάγνερ ε, ένα θέμα ήταν η διαφάνεια. Το ερώτημα μου είναι γιατί δεν έχουμε διαφάνεια στι ε, εξαγωγέ διπλή χρήση. Το έχουμε στι εξαγωγέ όπλων. Έχουμε αναχώρα, έχουμε κατηγορίες, ε, ζητήματα αδειοδότησης, ε, άρνηση κτλ. Σε μεγάλο βαθμό λεπτομέρειες. Γιατί δεν έχουμε συγκεκριμένες ε, πληροφορίες για τα διπλής κρίσης. Για την άλλη η Μαρίτια Σχάκε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους τους ομιλητές που ήρθαν στο Κοινοβούλιο και μας διαφώτισαν. Μετά από έξι χρόνια πίεσης από πλευράς του Κοινοβουλίου έχει φτάσει η στιγμή και ε, πρέπει να δούμε το status quo που για όσους δεν παρακολουθούν το ε, ζήτημα καθημερινά οδηγεί στο να υποφέρουν άνθρωποι οι οποίοι επικρίνουν την κυβέρνησή του και αυτό σε κάποιε χώρε σημαίνει φυλακή, βασαριστήρια ή και χειρότερα. Νομίζω πως είναι απολύτω θεμητό να φροντίσουμε στοχευμένα να δούμε τα ζητήματα εκείνα που κατασκευάζονται στην Ευρώπη και κάθε μέρα γίνονται μικρότερα και φθηνότερα. Άκουσα λοιπόν κάποιε συμφωνίε ότι θα πρέπει να απαιτείται άδεια όταν υπάρχει μια θεμητή ανησυχία και τώρα το ερώτημα είναι τι, πότε είναι θεμητή. Το πρώτο ζήτημα λοιπόν που ήταν σαφές είναι αυτό των ορισμών. Τι είναι παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ποιες τεχνολογίες ε, καλύπτονται από αυτή την νομοθεσία και αν πρέπει να περιλαμβάνεται η τρομοκρατία. Υπάρχει λόγο νομίζω να ανησυχούμε για το ότι η πρόταση Κομισιόν δεν είναι ακριβή. Ε, άκουσα το ότι δεν θα πρέπει να περιληφθούν οι ανησυχίε ε, για την τρομοκρατία. Υπάρχει κάποιο τρόπο όμω να δούμε το θέμα των ανησυχιών για την ασφάλεια. Ε, υπάρχει η ανθρώπινη ασφάλεια, αλλά υπάρχει και ευρύτερη ασφάλεια, μια εμπορική αγορά η οποία θα επέτρεπε σε τρομοκρατικές οργανώσεις να αγοράσουν αυτά τα συστήματα. Υπάρχει λοιπόν ένας εναλλακτικό ορισμός ε, εάν δεν μιλάμε για ανησυχία για την τρομοκρατία δεύτερο θέμα. Σε ποιο επίπεδο πρέπει να το δούμε. Άκουσα ξεκάθαρα από την Digital Europe ότι πρέπει να υπάρχουν παγκόσμιες προδιαγραφές. Καλό θα ήταν αυτό, αλλά δεν ζούμε σε ιδεώδη κόσμο. Οπότε είναι σαφές ότι αν ακολουθούσαμε τον παγκόσμιο μέσο όρο, θα είχαμε βεβαίω έναν αγώνα προς ε, τα κάτω. Πρέπει να επιδιώξουμε υψηλότερες προδιαγραφές και να παίξει ηγετικό ρόλο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα τώρα για το θέμα των ερευνητών που δεν θα πρέπει να πληγούν ε, από αυτόν τον κανονισμό. Δηλαδή αν κάνουν hacking ε, ή δοκιμάζουν ε, να διεισδύσουν συστήματα για να δοκιμάσουν ακριβώς το λογισμικό. Δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να γράψουμε κάποια εξαίρεση για αυτούς. Π.χ. κάποιες εταιρείες, αν ε, οι ερευνητές τους ακριβώς κάνουν δοκιμές για να δημιουργήσουν καλύτερη κυβερνοασφάλεια, ίσως ε, μπορούμε να κάνουμε κάποια θετική εξαίρεση για αυτούς. Ε, δεύτερον, άκουσα πολλές ανησυχίες για τους ορισμούς που είναι ασαφείς για το λογισμικό hacking ή επιτήρησης. Ε, θα σας βοηθούσε αν εστιάζαμε στην εξαγωγή δεδομένων από συσκευές. Δηλαδή να μην καθορίσουμε τις τεχνολογίες που μπορούν να μπουν στα τηλέφωνα του κόσμου ή τους υπολογιστές, αλλά να αρχίσουμε να, ε, να μιλάμε απλά για την ε, ανάστηση πληροφοριών από αυτούς τους υπολογιστές χωρίς ε, γνώση και συνένεση των χρηστών. Να εστιάσουμε δηλαδή στις δυνατότητες αυτών των συστημάτων. Μήπως αυτός ήταν καλύτερος ορισμός. Συγκεκριμένο ερώτημα στην Digital Europe. Πόσοι άνθρωποι εργάζονται ε, στα, μεταξύ, μέλη σας για τον έλεγχο των εξαγωγών χωρίς την τωρινή ενημέρωση και τέλος ποια είναι η χειρότερη κύρωση που υπάρχει αν μια ευρωπαϊκή εταιρεία κάνει εξαγωγέ χωρί την κατάλληλη άδεια. Τι είναι το χειρότερο που μπορεί να πάθει μια εταιρεία εάν δεν ζητήσει άδεια εξαγωγής σε χώρες που απαγορεύει ο ΙΕ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Βασενάρ κλπ. Ευχαριστώ, Μαρίμανε, για την ΚΟΕ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε μία συγκεκριμένη ερώτηση. Μετά από την παρατήρηση του κυρίου Βάγνερ, ο οποίος είπε ότι ο κόσμος ο οποίος ε, διαμαρτύρεται κατά του ελευθέρου εμπορίου δεν στηρίζει τις αξίες του ελευθέρου εμπορίου. Ίσως να μην κατάλαβα. Μου φαίνεται λίγο περίεργη αυτή η δήλωση και θα ήθελα να εξηγήσει τι εννοείται. Δηλαδή ποιες είναι οι αξίες του ελευθέρου εμπορίου, τι εννοείται ότι δεν στηρίζουν τις αξίες και τι ε, σημαίνει αυτό. Ενώ του ξέρετε αυτού του ανθρώπου, εγώ έχω διαδηλώσει πολλέ φορέ μαζί του και δεν έχω δει κάποιον ο οποίο ήταν κατά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή κατά τη προστασία του περιβάλλοντο ή κατά τη διαφάνεια. Δεν ξέρω δηλαδή τι Εννοείται ακριβώς με αυτή σα ε, την δήλωση, αν είναι το πρόβλημα με τις αξίες ή με τους ανθρώπους. Ευχαριστώ. Η κυρία Μπεγκίν για την EFTD. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να κάνω ερωτήσεις που εντάσσονται στην πραγματικότητα της βιομηχανίας και των επιχειρήσεων. Ίσως ε, πιο πολύ προς τον εκπρόσωπο της Digital Europe, αλλά όλοι μπορείτε να απαντήσετε αν θέλετε. Είναι δυνατόν να δοθεί απόκριση σε άδεια για εξαγωγή στα κράτη-μέλη εάν θεωρούσαμε ότι ο κανονισμός μπορεί να ισχύει αμέσως. Επίσης, το επιπλέον κόστος, αν εφαρμοστεί ο κανονισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα των ψηφιακών τεχνολογιών, πόσο θα μπορούσε να είναι. Η αύξηση τιμής ε, για τα μεμονωμένα προϊόντα δηλαδή. Και επίσης, θα ήθελα να καταλάβω, εάν κατά την άποψή σας ευσταθούν οι ευθύνε, η, κατανομή των ευθυνών μεταξύ των επιχειρήσεων και των ε, δημόσιων αρχών, όπως προκύπτουν από τον κανονισμό. Η ισορροπία που προβλέπει ο κανονισμός είναι αρκετή. Μήπως πρέπει να ελαφρύνει κάπως το γραφειοκρατικό άχθος που βαραίνει τώρα τις επιχειρήσεις. Ευχαριστώ. Μάλιστα, για τις απαντήσεις τρία λεπτά. Κύριε Βάγκνερ. Ευχαριστώ για την τεράστια αυτή πρόκληση. Θα κάνω ό,τι μπορώ. Να απαντήσω κοιτώντα προς τα πίσω. Και ανάποδα. Προς την κυρία Μινέρ, γιατί για προς την κυρία Βαγκίνη δεν νομίζω ότι έχω να πω εγώ κάτι. Για όσου βγήκαν και διαμαρτυρήθηκαν στου δρόμου για την εμπορική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Διαμαρτυρήθηκαν διότι θεωρούν ότι το εμπόριο όπω γίνεται δεν γίνεται για αυτού. Η πίστη και η ελπίδα του είναι ότι αν η μεταρρύθμιση τη διπλή χρήση προχωρήσει, θα μπορούσε η αξία του, η αλλαγή ανταλλαγή αυτών των προϊόντων θα μπορούσε εντασσόμενη στην ευρωπαϊκή πολιτική να αυξήσει και την πεποίθηση των ανθρώπων να θα ωφεληθούν από αυτή την εμπορική πολιτική. Δεν είναι δηλαδή άσκηση κριτική κατά των ε, ε, διαδηλωτών, αλλά θα υπάρξει περισσότερη πίστη εκτό ε, του σώματο αυτού, του θεσμικού αυτού οργάνου, από τον κόσμο. Βεβαίω, σε κάθε περίπτωση ο κόσμο έχει δικαίωμα να πει στου δρόμου να διαμαρτυρηθεί εφόσον θέλει. Για τι παρατηρήσει τη κυρία Χάκε, θα πρέπει να τα έχουμε λίγο κατά νου όταν μιλάμε για την εκμετάλλευση των συσκευών. Δεν είμαι βέβαιος ότι αυτή θα είναι η βέλτιστη λύση, αλλά σίγουρα είναι καλύτερη σε σχέση με αυτή που τώρα έχουμε. Θα πρέπει η συγκατάθεση των χρηστών και ο έλεγχος χρήσης των συσκευών είναι πολύ σαφής. Το να χάνουν τον έλεγχο των συσκευών τους οι χρήστες είναι σίγουρα τεράστια πρόκληση για την ειρήνη και την ασφάλεια στον κόσμο η ευθύνη ελέγχου μια συσκευή φαίνεται σε ατομικό επίπεδο πολύ μικρό, πολύ ίσονο σημασία θέμα, όμω πολύ γρήγορα μπορεί να πάρει τεράστιε διαστάσει. Οπότε αυτό που είπατε ήταν πολύ ενδιαφέρον και πολύ κέριο. Το ίδιο και για τι προτροπέ να βεβαιωθούμε ότι οι ερευνητέ κάνουν την ερευνά τους και με κάποιε εξαιρέσει μπορούν να προστατεύσουν την ακαιρεότητα αυτή τη έρευνα ακριβώ. Βεβαίω η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται αυστηρά πρότυπα. Αυτό είναι ανδιαφεσβήτητο. Όμω, όντω δεν μιλάμε εδώ για κανέναν αγγελικό κόσμο. Τα κράτη-μέλη κάνουν ε, μεμονωμένε προσπάθειε για να βρεθούν διευθετήσει για τα θέματα αυτά. Δηλαδή, αν περάσει αυτή η μεταρρύθμιση, θα έχουμε περισσότερο ίσου κανόνε παιχνιδιού, όχι λιγότερο. Για τη διαφάνεια, ερώτηση του κυρίου Λάγκε. Δεν υπάρχει για την ώρα σε αυτόν τον τομέα και πολλοί επισημαίνουν ότι οι εταιρείε δεν είναι πρόθυμες να ανοίξουν τα κοιτάπια τους εδώ. Αυτό ισχύει στην περίπτωση που τα άτομα οι πολίτες απευθυνθούν στις αρχές όπου υποχρεούνται να επιδώσουν κάποια έγγραφα αλλά δεν τα δημοσιεύουν στο, ε, ίντερνετ. Και τελευταία παρατήρηση για τις ρήτρες κάτσολ και αν μπορούν όντω να φέρουν αποτέλεσμα. Ήδη πολλές ρήτρες τέτοιου τύπου τις εφαρμόζουμε. Μπορούν να υπάρχουν, απλώς χρειάζεται σαφήνεια και βεβαιότητα για αυτές. Οι ρήτρες κάτσολ ε, εφαρμόζονται, είναι παράταση κάποιων πραγμάτων που ήδη εφαρμόζονται. Αυτή τη στιγμή θα μπορούσε να προκύψει απόκληση μεταξύ το ότι ένας εξαγωγέας θα πει σε μια διοδοτούσα αρχή από τη μια και στις εκθέσεις CSR από την άλλη. Αυτό δημιουργεί μια κατάσταση αντιφατική. Καλό θα ήταν να βεβαιωθούμε ότι αν έχει κανείς βέβαιη γνώση ε, ενός εγγράφου θα πρέπει να το μάθει και η άλλη αρχή, η, αδο, η αδειοδοτούσα κυρίως. Αυτός είναι ο σκοπός ε, των ρήτρων κάτσων. Κύριε Φιέγνερ, σας λείψαν κάποιες ναι, για τα κάτσολ, ε, για τις ρήτρες κάτσολ. Πέραν της εποπτείας της τεχνολογίας όμως, δεν ήταν μόνο αυτός ο στόχος και άκουσα πολλά σχόλια για τεχνολογία και το καθεξής. Εκεί ήθελα εγώ να σταθώ. Θέλετε να απαντήσω. Με συγχωρείτε. Προσπαθούσα να παραμείνω στο τρίλεπτο. Και κοίταζα τις ερωτήσεις που είχα ήδη σημειώσει. Ναι, είναι λογική η ερώτηση, αλλά είναι πολύ δύσκολο να απαντηθεί σε αυτό το πλαίσιο. Αν με ρωτάτε αν υπάρχουν ε, κλάδοι πέραν τη υποπτία ε, ή των ε, τεχνολογιών παρακολούθηση των συσκευών που αυτό είναι δυνατό, σαφώ. Αλλά ω εμπειρογνώμων δεν μπορώ να αρχίσω να σα δίνω παραδείγματα του ποδαριού. Θα έπρεπε να έχουμε μια καλύτερη κάλυψη του θέματος. Η Λούση. Ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να μην ξεπεράσω τα τρία λεπτά. Σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα να εμπλέξουμε την οργανωμένη κοινωνία των πολιτών. Ένα από τα βασικά που ανέφερα ήταν η έννοια ενό ετήσιου φόρουμ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποχρεωθεί να λάβει υπόψη τα αποδεκτικά στοιχεία που κομίζει η οργανωμένη κοινωνία των πολιτών. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για μας, να έχουμε μια λεωφόρο που θα βαδίσουμε ένα μέρος, ένα βήμα για να παρουσιάσουμε τα στοιχήματα τα στοιχεία μας από το να προσπαθούμε να ε, στριμώξουμε κάποιον ευρωβουλευτή τέτα τέτ για να συναντηθούμε μαζί του και να τον ενημερώσουμε συνέχεια. Αυτό ε, συμπεριλαμβάνει τη συνεισφορά της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών, θα δώσει φωνή στην κοινωνία και θα μας κάνει να υπάρχουμε και επισήμως. Έρχομαι τώρα στον κύριο Φιέλνερ. Σας ευχαριστώ. Δεν μας κουράζετε καθόλου με τις ερωτήσεις σας, αλλά ούτε και μας ρίχνετε στα μαλακά. Σημαντικό είναι να δείχνουμε περιπτώσεις που δεν καταστρατηγούν, δεν διευκολύνουν ε, τις καταστρατηγίες ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για παράδειγμα, το encryption, η κρυπτογράφηση. Υπάρχουν πολλές χρήσεις. Το θέμα είναι η διτή χρήση. Δηλαδή, Όλο αυτό το λογισμικό και υλικό που δημιουργείται μπορεί να έχει πάρα πολλές θεμητές χρήσεις. Δεν ρυθμίζουμε μόνο τους ηλέκτες που λένε ότι μπορούν να καταγράψουν οποιαδήποτε συνομιλία σε ακτίνα 2 χιλιόμετρων ή να διατηρήσουμε κάτι για την Τουρκία, για τον οποιοδήποτε άλλο για πέντε χρόνια. Μιλούμε για τεχνολογία που φτιάχτηκε κατάφορα με πρόθεση να ε, πλήξει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εμείς μιλούμε για τεχνολογία που δεν επινοήθηκε για αυτόν τον λόγο, αλλά τελικά καταλήγει να χρησιμοποιείται έτσι. Και ευχαρίστω να σας δώσω και περισσότερες λεπτομέρειες. Για την τροποκρατία δεν κατάλαβα πολύ καλά ποιο ήταν το ερώτημά σας να μου το ξαναθέσετε για να το ξανασκεφτώ να σας απαντήσω παρακαλώ στην κυρία ε, Σάκε ε, ε, για την έρευνα για θέματα ασφαλείας και τη δοκιμασία της, της δοκιμές στη διείσδυση, penetration και ούτω καθεξής, θα πρέπει να υπάρχει ένα είδος ανείχνευση, ηχνηλασιμότητα. Να μην κάνουμε την ερευνητική βιομηχανία να γονατίσει, όμως να φτάσουμε τελικά επιτόπου να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που προσπαθούν να δείξουν τις ευαισθησίες, την τροτότητα, την ευαλωτότητα των συστημάτων τεχνολογίας. Και για στην κυρία Μπεγκίν, αν πρόφερω καλά το όνομά σας, να σας μιλήσω για την ισορροπία μεταξύ εταιριών και ανάγκης ε, κρατικής ρύθμισης νομοθετικής. Ναι, πρέπει να ασκήσουμε ποιήση. Δίνεται έμφαση στην αυτορύθμιση, παρόλο που δεν αναφέρεται ξεκάθαρα. Καταλαβαίνω ότι οι αρχές αδειοδότησης έχουν συγκεκριμένη ροή εργασίας και έχουν φόρτο εργασίας, αλλά είναι σημαντικό το κράτος να μπορεί να πει ότι το τάδε πράγμα δεν είναι αποτελεσματικό και δεν συνάδει με τις διεθνείς μας υποχρεώσεις βάσει διεθνούς δικαίου. Αυτά προς το παρόν. Ευχαριστώ να επανέλθω με απαντήσεις. Ο Μάγνος. Ε, συγγνώμη, χρειάστηκα λίγη βοήθεια για να βρω το κουμπί του μικροφόνου. Να ερμηνεύσω το ερώτημα του κυρίου Μπούκνερ. Πώς συλλαμβάνεις και πιάνεις ένα κινούμενο στόχο. Όντως είναι, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και αυτή είναι και η πρόκληση. Το catch all όμως, οι ρήτρε ε, αυτές είναι μόνο σε WMD και τώρα προσπαθούμε να περιλάβουμε προϊόντα που είναι για αστική χρήση, που χρησιμοποιούνται από τους πολίτες. Έχουμε 1,8 εκατομμύρια προϊόντα. Χρειαζόμαστε σαφείς τεχνικές προδιαγραφές για να έχουμε catch-all, ε, ε, πλήρη σύλληψη για όλα αυτά τα προϊόντα. Αν μπορούμε όλα αυτά να τα βάλουμε στα συστήματα για αυτόματους ελέγχους, ε, τότε πρέπει να έχουμε πολύ σαφείς τεχνικές προδιαγραφές. Υπάρχει ανάγκη να αναθεώρησης πάρα πολλών ε, ε, αντικειμένων που βρίσκονται στον κατάλογο και αυτό δεν είναι καθόλου ρεαλιστικό ούτε πρακτικό. Θα είναι εξαιρετικά δύσκολο για εμάς παρόλο που είναι για έναν ανώτερο ευγενή σκοπό. Αυτά καταρχάς. Δεύτερο, για τον κύριο Φιέλτερ. Μελετάτε την κρυπτογράφηση και λέτε να μην διευκολύνουν, αλλά και η κρυπτογράφηση διευκολύνει. Οτιδήποτε μπορεί να διευκολύνει και τα ανθρώπινα δικαιώματα από τη μία και τα την τρομοκρατία από την άλλη. Εξού και είναι, σημαντικό να συλληφθεί με σωστό τρόπο για να ξέρουμε τι πρέπει να διαχειριστούμε και να διοικήσουμε στην βιομηχανία. Govern. Ηρωνικά, ε, αυτό που μας ε, έπληξε ήταν το λογισμικό για εισβολές, intrusion software. Έπρεπε εμείς να κάνουμε capture σε πάρα πολλές τεχνολογίες. Ε, πάρα πολλές καλές φιλοδοξίες έχουμε να ελέγξουμε τα πράγματα, αλλά είναι πολύ εύκολο να εκτροχιαστούν τα πράγματα και να χρειαστούμε εμείς οι ίδιοι capture technology. Άρα να προχωρήσουμε με πιο αργά βήματα. Τώρα, αγώνας προς τα κάτω για το ποιος θα είναι ο πιο βραδύς στην αντίδρασή του. Όχι, απαντώ, όχι δεν είναι το μόνο εργαλείο αυτό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βελτιώσει την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σε κάθε περίπτωση στην παγκόσμια κοινότητα μπορούν να βελτιωθούν οι έλεγχοι στις εξαγωγές. Ως Επιτροπή ε, έχουμε τη σχετική Επιτροπή που προσπάθησε να βρει ποιες είναι οι χειρότερες χώρες, προσπάθησε να συμπεριλάβει νέους ελέγχους στο πλαίσιο Βάσεναρ. Υπάρχουν εργαλεία και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αυξηθεί η προστασία ως προς τον αριθμό των απασχολούμενων, η εταιρεία μου απασχολεί 150 ανθρώπους στη συμμόρφωση για τις εξαγωγές και αν δεν πάρουμε άδεια, δεν είναι το πρόβλημα οι ποινέ που είναι σχετικά χαμηλέ και οι κυρώσει. Ενώ στι ΗΠΑ ο ανταγωνιστή μου χρειάζεται να πληρώσει 1,2 δι δολάρια το χειρότερο για μας είναι να μην αδειοδοτηθούμε πλέον, αν δεν συμπεριφερθούμε δεόντως και δεν βελτιώσουμε τη συμπεριφορά μας. Αυτό αρκεί για να συμμορφωθούμε το ότι δεν θα πάρουμε άδεια. Και ο χρόνος για την αδειοδότηση είναι από 40 έως 60 μέρες θα έλεγα. Το σύστημα αξιολόγηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι το πιο δύσκολο που μπορεί να γίνει. Άρα ε, η περίοδος 40-60 ημερών μπορεί να αυξηθεί. Εμείς είμαστε 150 άνθρωποι στην εταιρεία μου και στην Ιταλία. Οι Σουηδικές αρχές έχουν 22, στην Εσθονία είστε 5, τρεις ήσασταν πριν από λίγα χρόνια. Δεν είναι εύκολο το καθήκον, είναι μια ολοκληρή σειρά ελέγχων και σας ζητούμε να το εξετάσετε με ρεαλισμό. Ευχαριστώ. Η Λούση θέλει να παρέμβει, παρακαλώ. Θα είμαι εξαιρετικά σύντομη. Θα ότι δεν συμφωνώ με το υπονοούμενο ότι η κρυπτογράφηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επιθέσεις. Καταλαβαίνω ότι ως εργαλείο ασφαλείας εμποδίζει κάποια πράγματα, αλλά αυτό είναι το ίδιο επιχείρημα που θα ακούμε σε λίγα χρόνια ότι το firewall ή το antivirus ε, δεν είναι καλό γιατί έχει malware ε, το κράτος και εγώ τους εμποδίζω. Ευχαρίστω να το συζητήσω, αλλά διαφωνώ. Μάλιστα, Μαρίτια, θα ήθελα να κάνω μια... να ζητήσω από την ε, Digital Europe αν μπορεί να μου πει πόσοι εργάζονται ε, πάνω στο θέμα των ελέγχων εξαγωγών. Πρέπει να είναι χιλιάδες, ε. Α, κοίταξε, είμαι εγώ και η ομάδα μου. Αυτό ήταν ε, το ερώτημα. Το ένα που αφορούσε την πρόκληση και τώρα περνάμε στην πρακτική σκοπιά πώς θα γίνει το σύστημα πιο αποτελεσματικό. Και ο πρώτος ειδικό εδώ είναι πραγματικά από την σκοπιά της ε, πρακτικής, από την αρμόδια υπηρεσία για τον εξαγωγικό έλεγχο όπλων. Ο κύριος Πιέτς, έχετε τον λόγο. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Θα ήθελα να κάνω δύο παρατηρήσεις. Η υπηρεσία μας είναι η κεντρική αρχή αδειοδότηση στην Γερμανία για τα είδη διπλής ε, χρήσης. Είχαμε το 2010 πάνω από 10.000 τέτοιες αδειοδοτήσεις και αυξάνεται ο αριθμός των ειδών που υπάγονται στον ε, κανονισμό διπλής χρήση και σιγά σιγά αν συνεχιστεί αυτή η τάση θα φτάσουμε στις μισές σχεδόν εξαγωγές της ε, Γερμανίας. Και βεβαίω ε, βλέπετε τον όγκο της εργασίας μας. Δεύτερον, για μια δημόσια αρχή, όπως και για τις επιχειρήσεις, αποφασιστικό είναι ακριβώς, όπως υπόθηκε, ο Ευρωπαίος νομοθέτης να διατυπώνει τα πράγματα με σαφήνεια και ακρίβεια για να υπάρχει ακριβώς μια ασφάλεια προγραμματισμού σε επιχειρήσεις. Σκεφτείτε επίσης πως η παραβίαση αυτού του κανονισμού σημαίνει πως ε, θα πρέπει να, ότι δηλαδή όταν είχε γνώση ε, του τι πράττει μια εταιρεία σημαίνει ότι πλέον ε, αυτές οι πράξεις είναι ποινικά κολάσιμες. Μετά, επί της ουσίας, ε, τρία πράγματα. Το πρώτο αφορά τα αγαθά τα οποία σχετίζονται με παραβιάσεις ανθρωπίνων ε, δικαιωμάτων. Εδώ πέρα λοιπόν στην πρώτη πρόταση υπάρχει μια λίστα Ευρωπαϊκής Ένωσης για αγαθά διπλής χρήσης. Εδώ πέρα βλέπουμε από την πράξη την εισαγωγή μιας λίστας Ευρωπαϊκής Ένωσης μια τέτοια αγαθά πάρα πολύ θετικά. Θα πρέπει βεβαίως να περιοριστεί στο θέμα της τεχνολογίας και όχι στο ζήτημα των όπλων και του εξοπλισμού. Πρέπει να υπάρξει ξεκάθαρος διαχωρισμός μόνο. Λοιπόν, εάν δεν ε, πετύχει αυτό το διεθνές ε, κάθεστος, θα πρέπει να μιλήσουμε για αγαθά ε, τεχνολογικά στο παραδειγμα ένα 1β το οποίο τα οποία μπορούν να βοηθήσουν σε παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επίσης υπάρχει μια ομάδα ειδικών για την τεχνολογία επιτήρησης ε, που στην ε, Γερμανία κατέληξε το 2015 σε μια δική της θέση για τα είδη Βάσεναρ. Αναγκαίο επίσης είναι να έχουμε κάποιες παραμέτρους όταν μιλάμε για το διεθνές ε, καθεστώς και εδώ πέρα υπάρχουν κριτήρια πότε ένα αγαθό υπάγεται σε ένα καθεστώς ή όχι και η τωρινή πρόταση με το άρθρο 16 παραγραφός 2 προβλέπει ότι ε, για την ώρα δεν υπάρχει κάποιος ξεκάθαρος διαχωρισμός, δεν είναι αρκετά ακριβής η ορισμοί, οπότε εμείς είμαστε υπέρ ενός ξεκάθαρου παραρτήματος 1β, το οποίο θα αναγράφει όλα τα αγαθά αυτά, αλλά θα υπάρχει και ένας ξεκάθαρος ορισμός του πότε θα μπαίνει ένα αγαθό σε αυτή τη κλίση. Το δεύτερο θέμα το οποίο συζητιέται είναι η διάταξη catch all για τα ανθρώπινα δικαιώματα, μια γενική διάταξη. Οι γενικές προτινόμενες διατυπώσεις είναι πάρα πολύ γενικές από την σκοπιά της πρακτικής, δεν έχουν ξεκαθαρίσει ε, σημαντικά πράγματα. Παραδείγματο χάρη είναι η αιτιώδη σχέση η οποία απαιτείται με την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τι θεωρούμε βαριά παραβίαση που αναφέρθηκε και μη βαριά παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ποιε εθνικέ ή διεθνείς αρχές θα πρέπει να κάνουν αυτή την διαπίστωση και πώς θα τα ξέρει αυτά μια επιχείρηση. Επίσης βλέπουμε πως υπάρχει εδώ πέρα ο κίνδυνος ε, μιας τεράστιας γραφειοκρατίας η οποία θα διηγήσει σε αβεβαιότητα και θα εμποδίσει πολλές επιχειρήσεις να δραστηριοποιηθούν. Επίσης ε, δεν θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρξει αυτή η μεγάλη διακρατική διαβούλευση σύμφωνα με το άρθρο 4. Εμάς η λύση μας είναι για μια προσαρμογή του άρθρου 8 και 13 θεωρούμε ότι είναι η καταλληλότερη λύση για να μπορούμε να αντιδρούμε γρήγορα και με ευελιξία. Επίσης, ε, το άρθρο 4 παράγραφος 2 και σχετική ε, ρύθμιση που μιλάει για μια δέουσα επιμέλεια θα πρέπει νομίζω να ερμηνευτεί κάπως διαφορετικά. Είναι, πηγαίνει κάπως ε, πάρα πολύ μακριά. Και οι διατάξει οι οποίες υπάρχουν αυτή τη στιγμή θα πρέπει να έχουν τελείως διαφορετικέ προαπαιτούμενα Τρίτο θέμα, catch all για την τρομοκρατία. Εδώ πέρα έχουμε τις ίδιες επιφυλάξεις που ανέφερα και στα ανθρώπινα δικαιώματα. Κυρίως θεωρούμε πως ε, παραδόσεις ε, στα άτομα τα οποία συνδέονται με την τρομοκρατική προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, δεν μιλάμε για κάποια αγαθά. Εδώ πέρα καλύπτονται δυνητικά όλα τα αγαθά και θεωρούμε πως οι φυστάμενες διατάξεις είναι επαρκείς. Ε, δεύτερον, δεύτερο σύμπλεγμα διατάξεων, επέκταση του παιδιοφαρμογής και εδώ πέρα βλέπουμε μια προσθήκη του άρθρου 4 Β και ε, Δ ως υπερβολική δεν θεωρούμε ότι θα πρέπει να στοχεύσουμε σε κάτι τέτοιο. Αυτό μπορεί να γίνει κατά τη στιγμή της εξαγωγής, αλλά για έρευνες νομίζω ότι είμαστε σε λάθος διεύθυνση. Για την τεχνολογική υποστήριξη βλέπω πάρα πολλές θετικές ε, προσεγγίσεις στην πρόταση της Κομισιόν. Βεβαίω χρειάζονται εδώ πέρα διευκρινήσεις τι εννοούμε. Public domain ε, και έρευνα. Υπάρχουν βεβαίως ε, σε διεθνείς διατάξεις κάποιοι ορισμοί, αλλά θα πρέπει να δούμε και ποιες θα είναι και οι τεχνολογικές εξελίξεις, να υπάρξει κάποια ενημέρωση ή αναβάθμιση προϊόντων ε, τα οποία έχουν ήδη πολιθεί, κάτι τέτοιο θα μπορούσε να καλύπτεται ε, ίσως από την υποχρέωση άδεια. Χρειάζεται λοιπόν εδώ πέρα μια αξιολόγηση ίσως. Το επόμενο για τα έγγραφα 5 και 6 απαιτείται μεγάλη συζήτηση για διοικητικούς κανόνες όπως το θέμα της ε, διάρκειας της άδεια για την παγκόσμια και τη συνολική αδειοδότηση, υπό ποιε προϋποθέσεις ε, θεωρούμε πως ε, δεν είναι λογικό να υπάρχει μία και παγκόσμια αδειοδότηση. Επίσης, στις συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου βλέπουμε πως μία γενική άδεια ε, δεν ε, ε, είναι δυνατόν να συνεχίσει να υπάρχει στο υφιστάμενο status quo. Επίσης υπάρχουν και πολλά τεχνικά ζητήματα τα οποία μπορώ ευχαριστώ, να αναφέρω λεπτομερώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε. Τώρα θα δώσω τον λόγο την Αντέλα Διακονή, την Διευθύντρια της Φίλιψη για τον εξαγωγικό έλεγχο. Ευχαριστώ εκπρόσωπο και τους εποπτές ε, της Ολλανδίας, όχι μόνο την Philips. Η προτινόμενη μεταρρύθμιση της διπλής χρήσης είναι κάτι που στηρίζουν οι επιχειρήσεις με τον εξυγχρονισμό του ρυθμιστικού πλαισίου για τη διπλή χρήση. Διότι θα πρέπει και αποτελεσματικά να διαχειριστούμε τις αναδυόμενες απειλές, αλλά μην το ξεχνάτε και τις ευκαιρίε να περτιώσουμε τις ζωές των ανθρώπων. Γι' αυτό εμπορευόμαστε. Όχι μόνο για να γινόμαστε καλύτεροι, αλλά για να βελτιώσουμε και τη ζωή των ανθρώπων. Ο εξυγχρονισμό πάντω, όπω και η κοινοτομία, εγκυμονούν ε, σοβαρέ ευθύνε για του νομοθέτε. Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι υπάρχει νομική βεβαιότητα. Ότι υπάρχει σαφή νομική γλώσσα και αντιμετωπίζονται οι σοβαρότερε μέρημνε. Η βασική μα ανησυχία στι εταιρείε όπω η Philips είναι τα ε, πλεονεκτήματά μα από ανταγωνιστική σκοπιά και η νομική βεβαιότητα. Για να το πω πολύ ξεκάθαρα, εάν δεν κάνουμε σωστή μεταρρύθμιση για τα επόμενα 10 χρόνια, δεν θα, όχι απλώς δεν θα πετύχουμε τους στόχους ασφάλειας, αλλά τις ευρωπαϊκές εταιρείες θα τις κάνουμε να πτωχεύσουν, θα φαλήρουν ή θα φύγουν από την Ευρώπη. Δύο βασικά κριτήρια για την επιτυχία λοιπόν που θεωρώ ότι θα έπρεπε να έχει μεταρρύθμιση. Για να είναι τα συστήματα ελέγχου ε, θωρακισμένα και για το μέλλον. Προέκυψαν για τα λόγια κάποιων από του ομιλητέ αλλά και του εκπροσώπου τη Μπάρτα. Να θυμηθούμε το άρθρο 3 τη συνθήκη για την λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση να συμβάλλει στην ειρήνη και την ασφάλεια, αλλά και την, το ελεύθερο και δίκαιο εμπόριο και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ναι, νομίζω το να βρούμε το σωστό σημείο ισορροπία είναι ένα κριτήριο επιτυχία. Η θέση ε, της βιομηχανίας σε με την τωρινή πρόταση είναι λίγο επιφυλακτική διότι υπάρχουν κάποιε ανυπολόγιστε συνέπειε. Το δικαίωμα στην υγεία και το δικαίωμα στον ιδιωτικό βίολογο, χάρη. Το γεγονό ότι η τωρινή πρόταση μπορεί να καταλήξει να μην ε, επιτρέπει να επιτευχθούν αυτά. Γιατί, Γιατί η διτή χρήση τη τεχνολογία, η διπλή μάλλον χρήση τη τεχνολογία, αυτή που θέλουμε να ελέγχουμε, πολλέ φορέ μα προστατεύει. Προστατεύει και τα αρχεία μα, για να το πω έτσι. Οπότε οι ανησυχίες του κλάδου είναι ε, σοβαρές και ο τρόπος να μένουμε εκτεθειμένοι σε από τρομοκράτες, από οργανωμένα έγκλημα έρχεται από αλλού. Έτσι λοιπόν η μεταρρύθμιση αυτή μπορεί να γίνει ένα πολιτικό εργαλείο και γίνεται πολιτικού χαρακτήρα. Λόγω ακριβώς αυτού του πολιτικού χαρακτήρα δεν θα υπάρξει ποτέ πλήρης ευθυγράμμιση. Θα είναι δύσκολο αυστηροί έλεγχοι να εφαρμόζονται μέσα από ένα αυστηρά τεχνικό και τεχνολογικό εργαλείο όπως ο κανονισμός για τη διπλή ή τη διτή χρήση. Θα πρέπει λοιπόν εδώ να επικεντρωθούμε στον προτινόμενο μηχανισμό ελέγχου και για τις εταιρείε και για τον ρυθμιστή και να δούμε πώς είναι δυνατόν να παραταθεί το υπάρχον σύστημα και να είναι η έλεγχη αποτελεσματική, αλλά και να επιτρέπουν την επίτευξη των στόχων που θέλουμε. Αν υπάρχει ένα σαφή ορισμό που τον υποδέχονται όλοι, και οι εταιρείε και επιχειρήσει και οι νομοθέτε και οι εταιρείε εξαγωγέ, αλλά και όσοι προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μην ξεχνάμε, παραβίαση ανθρώπινα δικαιώματο για ένα κατό μέλο μπορεί να είναι κάτι το διαφορετικό από ότι για ένα άλλο. Και ακόμη και δύο άνθρωποι μπορεί να διαφωνούν στα πλαίσια μια συζήτηση. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Θα πρέπει να υπάρχει ένα κατάλογο χωρών που εμπίπτουν σε οποιαδήποτε από τι κατηγορίε που αναφέρεται στη νέα πρόταση, όπω οι μη ευαίσθητε χώρε οι ευαίσθητες χώρες, ε, το ε, απολυταρχικό καθεστώς, οι περιοχές, ε, οι διαφρονικούμενες συγκρούσεων. Αυτά είναι σοβαρή πολιτική τομή και θα πρέπει να δούμε γιατί η πολιτική διαδικασία θα μας επιτρέπει να πετυχαίνουμε την δέουσα επιμέλεια. Ναι, έχουμε πολύ δέουσα επιμέλεια σε επίπεδο και την παίρνουμε πολύ σοβαρά. Όμως, η έλεγχη των εξαγωγών απαιτούν να είμαστε πιο αντικειμενικοί. Και με την πρόταση για τι ρήτρε χατσόλου. Και επίση πρέπει να υπάρχει και σαφή ορισμό των παραμέτρων των τεχνολογικών που θέλουμε να έχουμε. Το ακούσατε και από την Business Europe και την Ericsson. 1,8 εκατομμύρια είδη προϊόντων προσπαθούν να ταξινομηθούν βάσει αυτών των τεχνικών ε, προδιαγραφών, όμω ε, δεν είναι εύκολο. Είναι σχεδόν αδύνατο να τα εντάξουμε κάπου. Είναι τεράστια πρόκληση για όλου του εμπρογνωμόνε του κλάδου. Η δική μου λοιπόν ε, η προτεραιότητα μαζί με τους νομοθότες, τους ρυθμιστές και τους ελεγκτές των εξαγωγών είναι εάν η πλήρης ευθυγράμμιση δεν μπορεί να εφαρμοστεί παράταση να υπάρξει. Ε, βέβαια λόγω πολιτικών αιτίων δεν πρέπει να ε, εφαρμόσουμε την πρόταση καλά και ντε, αλλά να δούμε πώς δεν θα δημιουργήσουμε περισσότερους φραγμούς, γιατί ε, ένας ελεύθερος κανονισμός δεν θα δώσει βεβαιότητα για το μέλλον. Επίσης, δεν μπορεί μονομερός η Ευρωπαϊκή Ένωση να ρυθμίσει ένα κατάλογο προϊόντων ε, υπό το τίτλο διπλή χρήση. Οι μονομερείς κατάλογοι είναι κάτι που θα πρέπει να το προσέξουμε. Γιατί, διότι εάν ξεφύγουμε από το πολυμερές καθεστώς και σύστημα, όχι μόνο νομικέ βέβαια το θα δημιουργήσουμε, αλλά και απογοητεύσει και το αποτέλεσμα θα είναι κατά τη γνώμη μου απλό. Θα στρεβλώσουμε τελείως τον ανταγωνισμό που ήδη τον έχουμε στον κυβερνοχώρο τη δηλαδή, δεν θα πετύχουμε τους στόχους των προϊόντων που θέλουμε μονομερώς να ελέγχουμε, θα κυκλοφορούν έτσι κι και θα είναι αντικείμενο εμπορία άλλων χωρών και οι κακοί πάλι θα καταφέρουν να προμηθευτούν αυτό που θέλουν, αλλά από κάπου αλλού. Θα πρέπει λοιπόν οι νομοθέτες να σκεφτούν το εξής μην επιμένετε να υπάρχει οπωσδήποτε, μάλλον να μην ξεχνάμε ότι μπορεί να υπάρχει ευθυγράμμιση με άλλα συστήματα εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση και να βασιζόμαστε στι τεχνικέ παραμέτρου των προϊόντων και όχι στι ενδεχόμενε κρίσει. Παράδειγμα, ένα φορείο νοσοκομείου μπορεί να χρησιμοποιηθεί και αυτόδητο. Δεν θέλω να επεκταθώ σε αυτό το παράδειγμα περαιτέρω, διότι δεν είναι αυτό το θέμα μας, αλλά και μια καταληκτή διαπραγμάτευση. Ε, Πιστευόμαστε του ρυθμιστέ και νομοθέτε ότι θα πετύχετε το καλύτερο δυνατό για τι επιχειρήσει, εταιρείε και το εμπόριο. Χρειάζεται νομική βεβαιότητα, σαφή, ξεκάθαρη ε, νομική γλώσσα, ε, ίσοι κανόνε, ισότιμοι κανόνε παιχνιδιού και ε, ξεκάθαρη στάση. Είμαστε πρόθυμοι ε, ως εταιρείε και ε, επιχειρήσεις να πετύχουμε τον ίδιο στόχο μαζί σας για το καλό των πολιτών και η έλεγχοι των εξαγωγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αποτελέσουν υπόδειγμα για τον υπόλοιπο κόσμο. Σας ευχαριστώ πολύ. Και περνάμε τώρα στο Μάλτε Πόλμαν, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ουτιμάκο GmbH. Σας ευχαριστώ πολύ. Εκτιμώ ιδιαίτερος την, την ε, δυνατότητα που δίνεται σε μια μεσαία επιχείρηση να απευθύνει ε, το λόγο στο ακροατήριό σας. Είμαστε από το Άχεν της Γερμανίας και θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε την πραγματικότητα από δικής μας πλευράς, να σας πούμε τι κάνουμε και πώς ε, ε αντιμετωπίζουμε τη διπλή χρήση. Εργαζόμαστε στον τομέα της κυβερνοασφάλειας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε περίπου 170 απασχολούμενους. Είμαστε σε ειδική, ε, ειδικό κατάλογο στη Γερμανία. Έχουμε καλή συνεργασία με τις γερμανικές αρχές, με την BAFA, BAFA. Δίνουμε κανόνες ασφαλείας, κυρίως από πλευράς φωτογραφικών προϊόντων σε διάφορες υποδομές και έχουμε τα ίδια προϊόντα σε πολλές και διαφορετικές εφαρμογές και χρήσεις. Εθνικές ταυτότητες για τη γερμανική κυβέρνηση, έλεγχος των ατόμων στο αεροδρόμιο Σίπχολ του Άμστερνταμ, έλεγχος πρόσβασης στο κτίριο Μπερλεμάν, ε, στις Βρυξέλλες, ε, τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου και άλλων για οχήματα διαφόρων αυτοκινητοβιομηχανιών. Έχουμε εγκαταστάσεις σε πάνω από 80 χώρες και Ασχολούμαστε πάρα πολύ και μας ενδιαφέρει η συμμόρφωση βεβαίως με, τις, με τα διαφορετικά καθεστώτα ελέγχου των εξαγωγών αναχώρα. χώρα. Τέθηκε, τέθηκε το ερώτημα ποια είναι η προσπάθεια που πρέπει να καταβάλει μια επιχείρηση για να είναι πραγματικά ηθική να σας δώσω την εικόνα που δείχνει την πραγματικότητά μας. Συμμόρφωση με OFAC και ESG ε, πάντοτε είναι υψηλή προτεραιότητα, δηλαδή συμμόρφωση για με τα ε, θέματα περιβάλλοντος, τα κοινωνικά και τα θέματα σωστής και χρηστής διακυβέρνησης και διαχείρισης και συμμόρφωση με τα OFAC. Έχουμε εσωτερικές διαδικασίες, διεργασίες, έχουμε θέσεις οργάνων στη διοίκηση ανθρώπων που ασχολούνται με αυτό, έχουμε και εξωτερικούς συνεργάτες και συμβούλους για που μας βοηθούν στη συμμόρφωση. Και επειδή εμείς προμηθεύουμε με κρίσιμη σημασία υποδομές, πρέπει να στοχεύουμε στο και το πράττουμε στο Know Your Customers Priority. Γνωρίζετε να γνωρίζουμε τις προτεραιότητες του πελάτη που είναι κράτη και μεγάλοι οργανισμοί οι πελάτες μας. Στόχος μας λοιπόν είναι αυτός δεν είναι κάτι που πάντοτε επιβάλλεται εύκολα σε μεγάλους εμπορικούς εταίρους και αναφέρομαι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο με τη ΣΥΠΑ και την Κίνα. Το να συμμορφωνόμαστε με τα προαπαιτούμενα είναι μεγάλη προσπάθεια για εμά και το πράττουμε. Έχει άμεσο αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητά μα, γιατί ανταγωνιζόμαστε με άλλου παρόχου κυβερνοασφάλειας που δραστηριοποιούνται στη Βόρεια Αμερική και στη Κίνα και πρέπει να συμπεριλάβουμε αυτό το κόστο στα συμβολέα μα και δεν ξέρω κατά πόσο είμαστε πάρα πολύ ανταγωνιστικοί. Το σημαντικό είναι να υπάρχει level playing field. Αυτό είναι καθοριστικό στο σημερινό κόσμο. Δεν ξέρω κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να το επιτύχει. Οι αρχές είναι η μπάφα γιατί το 99% των εξαγωγών μας πάει μέσα από τη γερμανική θηγατρική και το USUK και τη θηγατρική στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο. Θέλουμε να έχουμε ένα καθεστώς επιχειρηματικής ασφάλειας και να μπορούμε να δραστηριοποιηθούμε με σιγουριά για το ότι δεν θα αλλάζει το πλαίσιο κάθε τρεις και λίγο. Έχουμε ε, εξωτερικές αξιολόγησεις της συμμόρφωσής μας και της δέουσας επιμέλειας σε ε, πολύ τακτά χρονικά διαστήματα. Η τελευταία ήταν με το BSR, εμπειρογνώμονες μη κυβερνητική οργάνωση που εδράζεται στη Νέα Υόρκη. Όχι μόνο αρχές μας ελέγχουν για τη συμμόρφωσή μας, ούτε μόνο ε, κάθε αίτηση ξεχωριστά για συγκεκριμένη άδεια ελέγχεται για τη συμμόρφωση, αλλά είναι και ένα προαπαιτούμενο σύνηθες ε, να μας επιτερούν για τη διεργασία μας και κατά πόσο συμμορφωνόμαστε. Έχουμε χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τη Γερμανική Κρατική Τράπεζα Επενδύσεων ε, και έχουμε και επενδυτές με ίδια κεφάλαια από την EQT, ε, το, το μεγαλύτερο ταμείο και hedge fund με ίδια κεφάλαια επενδυτικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλοι αυτοί μας ζητούν να, να σεβόμαστε και να απαιτούν από εμά να τηρούμε τα προαπαιτούμενα και το πράττουμε. Έχω την αίσθηση ότι βεβαίως είναι και πολιτική αυτή η διαδικασία, αλλά ε, έχω την εντύπωση ότι τα σχόλια των εμπειρογνωμόνων δεν έχουν απεικονιστεί στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο βαθμό που θα θέλαμε. Ενδεχομένως αυτό και για λόγους πολιτικούς. Τώρα ε, τηρεί το ε, επιδιώκει το στόχο του και τον επιτυχάνει με ανάλογες προσπάθειες και όχι δυσανάλογες. Η απάντηση είναι ναι, αλλά ε, οι αιτήσει που υποβάλαμε στο παρελθόν χρειάζονταν πάρα πολύ χρόνο για να έχουμε απάντηση. όλες, όλα τα περισσότερα αιτήματα για διπλή χρήση έχουν να κάνουν με τον τομέα της κρυπτογράφησης. Ο τωρινός ορισμός της κυβερνοεποπτείας ε, θα αντέξει και στο μέλλον. Εγώ πιστεύω ότι σε λίγα χρόνια θα έχετε μπροστά σας ένα αντίστοιχο κείμενο και θα νιώθετε για το αντίστοιχο μελλοντικό κείμενο με το, τρο... το, με το δύο τρόπο με το οποίο νιώθετε τώρα για το κανονισμό για την κρυπτογράφηση. Δηλαδή, οι ορισμοί είναι έτσι διατυπωμένοι που επιφέρουν παράπλευρες απώλειες. Είναι πολύ αδύναμοι οι ορισμοί, πρέπει να γίνουν πολύ πιο σταθεροί, πολύ πιο στέρεοι και πολύ πιο σαφείς και ακριβείς. Ε, ιδαλλιώς θα υπάρξει ε, πρόβλημα και στο μέλλον. Τώρα, ε, είναι δύσκολο το θέμα της ε, ανθρώπινης ασφάλειας να καλυφθεί επαρκώς από όλα τα κατσόλ. Είναι δική μου ευθύνη ως το συμβούλου να έχουμε σωστή εικόνα εδώ. Έτσι όπως, η έτσι όπως έχει η πρόταση αυτή τη στιγμή, δεν βελτιώνει τη διαδικασία. Η προσέγγιση με βάση τη λίστα είναι κάτι που αυτόματα το κάνουμε ως εταιρεία. Τέσσερις-πέντε φορές τη μέρα κάνουμε τέτοιους ελέγχους. Ε, είναι μια διαδικασία που μπορεί κανείς να κάνει ε, χωρίς να απασχολήσει πάρα πολύ εργασιακό δυναμικό όταν είναι μια μεσαία επιχείρηση. Το catch all χρειάζεται πάρα πολλούς ανθρώπους. Είναι πάρα πολύ δυσχερές και η ασφάλεια για το επιχειρηματικό περιβάλλον είναι πολύ σημαντική στις διεθνείς συμφωνίες που συνάπτει μια ε, εταιρεία. Ε, όταν ακούω ότι έρχονται κατευθυντήριες γραμμές και θα επέλθουν είναι τεράστιο πρόβλημα για μια επιχείρηση γιατί εμείς δεν συνάπτουμε συμβόλαια με τους Ω μας ως προμηθευτές ε, τα μισά και το άλλο μισό συμβόλαιο να το υπογράψουμε του χρόνου. Ε, θα θέλαμε να υπάρχει εναρμονίση και συγκεκριμένα πράγματα. Και ο Μάγνος ανέφερε το το πόσο άνισα εξοπλισμένες είναι οι αρχές ελέγχου των διαδικασιών εξαγωγών από τη μία χώρα στην άλλη, ε, πρέπει τα πράγματα να γίνουν πιο ακριβή, πιο συγκεκριμένα, να μπορούν να λειτουργήσουν στην πράξη και ελπίζω και εύχομαι η διαδικασία εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμβάλλει στη βελτίωση της διατύπωσης του κειμένου. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε να σας απευθύνω το λόγο. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα έχουμε ερωτήσεις. Εισηγητής κ. Μπούχνερ. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα έχω μια ερώτηση στον κύριο Πίτση. Πώς ε, γίνεται, μας είπατε ότι θέλουμε να υπάρχει αξιοπιστία των ε, χι ε, ατόμων. Πώς εξηγείτε το ότι υπάρχουν ε, πολλές πολύ κρατικοί θεσμοί που είναι διεφθαρμένοι. Δηλαδή πουλάτε τα πράγματα σε κάποιον ο οποίος έχει στην αρχή καλές ε, προθέσεις ας πούμε και μετά υπάρχουν ε, π.χ. δωροδοκίες. Δεν είναι αδιανόητα πράγματα αυτά. Δηλαδή εγώ έχω κάποιες δυσκολίες με αυτά τα οποία μας λέτε. Το δεύτερο είναι μια απέτηση που αναφέρατε και οι δύο θέλετε μια λίστα ε, τεχνολογίας και όχι ε, σκοπού χρήσης. Απλό παράδειγμα. Η πλατεία της Ουράνιας Ειρήνης στο Βερολίνο 1989 η διαδήλωση κατεστάλλει με τεθωρακισμένα. Δύο χρόνια αργότερα, λίγα χρόνια αργότερα, 2009, διαμαρτυρίες ε, κατά της νοθείας ε, του Αχμαντίνετζάντ. Εκεί πέρα η εξέγερση κατεπνίγει πολύ πιο έξυπνα μέσω τεχνολογίας επιτήρησης. Εάν γινόταν κάτι τέτοιο πάλι σήμερα θα χρησιμοποιούνταν άλλη τεχνολογία, ξέρετε τι εννοώ νομίζω. Οπότε ε, αν περιοριστούμε λοιπόν σε συγκεκριμένη τεχνολογία ή συγκεκριμένα προϊόντα, απλά θα μας ξεπεράσει η εξέλιξη της τεχνολογίας. Τι άποψη έχετε. Και τέλος, αναφέρθηκε μια απόκληση από τις πολυμερείς λίστες. Κοιτάξτε, ε, κάποια συστήματα, η Βάσεναρ παραδείγματος χάρη, είναι πάρα πολύ αργά και η τεχνολογία εξελίσσεται πολύ πιο γρήγορα τι θα κάνουμε ο, αν ε, βασιστούμε σε τέτοιες άκαμπτες πολυμερείς λίστες. Σας ευχαριστώ για το ΕΛΚ ο κύριος Φιέλνερ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το πρώτο μου ερώτημα είναι για την κυρία Διακόνου. Ναι. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Αναφέρατε τρία προβλήματα, τρεις απειλές για τις αυτόνομες ε, λίστες. Και θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση, δεν ξέρω, ίσως είναι αδύνατη, ίσως όχι. Είναι κάτι το οποίο ε, θεωρείτε ότι ξέρετε ποιοι είναι οι κίνδυνοι, γιατί τώρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι ναι, οι αυτόνομες λίστες ε, είναι κάτι το νέο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ξέρουμε πως η Γαλλία και η Γερμανία έχουν ήδη ε, προχωρήσει πέρα από το Βασενάρ. Δηλαδή θα μπορούσατε ε, να δούμε κάποια από αυτά τα πράγματα τα οποία φοβάστε να συμβούν στη Γαλλία ή τη Γερμανία επειδή πήγαν παραπέρα και εξοπλίσαν κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να ονομάσουμε ξέρω, γερμανική ή γαλλική αυτόνομη λίστα. Δεύτερη ερώτηση, για να επανέλθω ίσως σε κάποια ερώτηση μιλάμε για catch-all και τα λοιπά. Και το αντιλαμβάνομαι, εντάξει. Αλλά διαβάζοντάς το αυτό, εγώ και ο κύριος Βάγνερ ε, έχουμε την εντύπωση ότι στη σημερινή πρόταση αφορά μόνο την επιτήρηση. αλλά δεν ισχύει αυτό. Ε, ξέρω πως η Κομισιόν λέει ότι είναι στοχευμένο, αλλά αφορά τα πάντα και ε, κύριε Πούλμαν, εάν ε, βεβαίω κάτι είναι πυρικά κολάσιμο, μπορεί να πάει κάποιο ε, στη φυλακή. Σημαντικό να ξέρουμε λοιπόν περί τίνο πρόκειται. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω, γνωρίζοντας ότι έχουμε μόνο την αξιολόγηση αντικτύπου για το κάτσολ, για την τεχνολογία κυβερνοεπιτήρησης, θεωρείτε ότι υπάρχει ανάγκη για κάτσολ πέρα από αυτόν τον τομέα. Γιατί δεν ξέρω, ίσως για να κοιμάται καλύτερα και όσο τα βράδια, καλό είναι νομίζω να σκεφτούμε τον ορισμό. Σας ευχαριστώ. Κύριε Πίτς. Ναι, ναι, αλλά είμαι σκιώδης εισηγητής για τους σοσιαλδημοκράτες, οπότε έτσι πάει η σειρά. Κύριε Πίτς. Αναφερθήκατε στην πρακτική στη Γερμανία. Αν το συγκρίνετε με την πρακτική σε άλλες χώρες της Ένωσης, υπάρχει διαφοροποίηση που θα μπορούσε ίσως να οδηγήσει στο ότι κάποιες επιχειρήσεις θα μπορούσαν να πάνε σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, τελικά ε, πώς πρέπει να γίνει ευρωπαϊκό το, το σύστημα. Ελπίζω να μην σα πάρει τη δουλειά καμία ευρωπαϊκή υπηρεσία και στον κύριο Πούλμαν. Ποια είναι τα κριτήρια για επένδυση. σε επενδύσεις, ε, παραδείγματος χάρη στην περίπτωση της Γερμανίας, είναι το εάν έχουν τα προσόντα οι εργαζόμενοι, είναι η υποδομή ή είναι όντως ζήτημα νομοθεσίας διπλής χρήσης. Αλέγατε πως ε, θα μπορούσε αυτό να οδηγήσει σε επένδυση και παραγωγή εκτός της Ένωσης. Και τώρα, αν είμαι Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Έχω δύο ερωτήσεις. Η πρώτη απευθύνεται στον κύριο Πίτς και στην κυρία Διακόνου. Ο κύριος Πίτς είπε πως κάποιοι κανόνες είναι πολύ επιβαρυντικοί για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και διέκρινε βαριές και μη παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και η κυρία Διακόνου είπε πως μπορεί να βλάψουν τις επιχειρήσεις κάτι τέτοια. Συμφωνώ μαζί σας πως υπάρχει κάποιο πεδίο έντασης μεταξύ καιροτομία, γραφειοκρατίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αλλά πρέπει να διαλέξουμε τι τελικά υπερισχύει. Εγώ ε, θα μπορούσα, δεν ξέρω, θα ήσασταν κι εσείς σε θέση να δεχτείτε λιγότερη καινοτομία και λιγότερα κέρδη μετά, κατόπιν. Είπατε ότι η εταιρεία σας ε, έδωσε στο καθιστός Ασάντ μια συσκευή παρακολούθησης υποκλοπών και υποκλοπών φαξ. Και οπωσδήποτε κάτι τέτοιο είναι μη επιθυμητό. Αλλά... Βλέπουμε εδώ πέρα λοιπόν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα προς αποφυγή. Πώς μπορούμε λοιπόν να αλλάξουμε το κανόνες για να αποφευθούν τέτοιες συμφωνίες δισεκατομμυρίων. Σας ευχαριστώ. Δίνω ξανά τον λόγο στους ειδικού για τρία λεπτά ο καθένας κύριε Πίτσου. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ξεκινήσω με την τελευταία ερώτηση. Στην πρόταση της Κομισιόν άρθρο 4 Δελτά αναφέρεται ρητός ότι αγαθά τα οποία δεν αναφέρονται ε, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για σοβαρές παραβιάσεις. Το σοβαρές παραβιάσεις είναι, είναι διατύπωση της ε, Κομισιόν. Και λέει ότι θα πρέπει η επιχείρηση να ενημερώνει τις αρχές όταν έχει γνώση για σοβαρή παραβίωση. Ε, ε Βεβαίω, πράγματι, εδώ πέρα είναι το ερώτημα τι γίνεται αν γνωρίζει ο πολιτής ότι πρόκειται για απλή ας πούμε παραβίαση και ποια είναι η σοβαρή και η απλή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν μπορώ και εγώ να... Είναι διαφορετικό θέμα, μπορεί να διαφέρει η άποψη στη Γερμανία από ό,τι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα για την ερώτηση πώς έχει η κατάσταση στα άλλα κράτη-μέλη. Ε, εδώ και 25 χρόνια δεν έχω δει κάποια επιχείρηση η οποία μόνο λόγω των εξαγωγικών ελέγχων μετέφερε την παραγωγή της από τη Γερμανία, ξέρω εγώ, στη Βρετανία ή τη ΣΥΠΑ. Είναι ε, πολλοί άλλοι λόγοι φορολογικοί και άλλοι που είναι πολύ πιο αποφασιστικοί από δύο-τρεις ε, απορρίψεις ε, της υπηρεσίας μας. Και επίσης προβλέπει ο κανονισμός πως αν κάποιο αγαθό βρίσκεται στη Γερμανία αλλά η εταιρεία στην ε, Γαλλία θα έπρεπε να μας ε, συμβουλευτούν οι Γάλλοι συνάδελφοι. Ε, ακριβώς για να αποφεύγουν αυτό το οποίο λέτε, δηλαδή να μεταφερθεί ολόκληρη η παραγωγή σε άλλη χώρα. Και μετά για τα θέματα του κυρίου Μπούχνερ, τι εννοούμε εδώ πέρα τρομοκρατία. Υπάρχει, υπάρχει νομίζω ένα Ευρωπαϊκό κανονισμό για το εμπάργκο που περιλαμβάνει νομικά και φυσικά πρόσωπα τα οποία έχει καθορίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ω ε, τρομοκράτε. Ε, σε αυτά έχει συμφωνήσει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι είναι τρομοκράτε. Τώρα το τι είναι τρομοκρατία είναι μια ακόμη ευρύτερη συζήτηση ακόμα και από το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και μετά πότε απαγορεύεται η μεταπόληση και αν πολιθεί κάτι 3, 4, πέντε φορές και πού θα καταλήξει στην αλυσίδα. Κοιτάξτε, ε, δεν το ξέρει η βιομηχανία και δεν το ξέρουμε και εμείς ως αρχή. Είναι πράγματι ένα πρόβλημα το οποίο ε, μόνο από την δυνατότητα μεταπόλησης ε, πρέπει να μας υποψιάσει. Επίσης, υπάρχει ακόμα ευρύτερο πεδίο εφαρμογής αν μιλάμε για πιθανότητα μεταπόλησης και όχι για σίγουρη χρήση. Και βεβαίως και αυτό είναι αιτία απόρριψης. Και έρχομαι εδώ πέρα σε ένα παράδειγμα με την ε, πλατεία της ε, Κίνας. Μα αν ξέρω εκ των προτέρων ότι θα πάει για καταπίεση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, υπάρχουν πολλές νομικές δυνατότητες και αν το ξέραμε εκ των προτέρων, θα έπρεπε, κατά την άποψή μου, να υπάρξει απαγόρευση. Αν μια επιχείρηση λέει ότι εγώ έχω θετική γνώση ότι το προϊόν μου θα χρησιμοποιηθεί 100% για βαριά παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ε, <laughs> δεν έχει να συζητήσουμε κάτι. Έτσι, ξεκάθαρη απαγόρευση. Αλλά η πιθανότητα δεν επαρκεί όμως. Και τέλος, πολυμερείς ε, λίστες. Ναι, είναι κάτι το δυσκίνητο Παραδείγματο χάρη, ε, μέχρι και σήμερα οι Αμερικανοί δεν ε, τις ε, εφαρμόζουν. Γι' αυτό οι Γερμανοί έχουν μια εθνική θέση. Είχαμε το τελευταίο έτος γύρω στις 20 εγκρίσεις και δύο απορρίψεις. Και οπότε σας είπα, καμία εταιρεία δεν έφυγε από τη Γερμανία για τον λόγο αυτό. Και πρόκειτο για πολιτικά προϊόντα. Γι' αυτό σας είπα, έχουμε κάνει μια εθνική λίστα και η θέση μας είναι νομίζω αρκετά ξεκάθαρη. Σας ευχαριστώ, Αντέλα. Θα προσπαθήσω να απαντήσω κατάλογος τεχνολογικών μέσων έναντι σκοπού. Νομίζω ότι ο κατάλογος της διπλής χρήσης θα εντοπίζεται στην πιθανή κακή χρήση κάποιων αγαθών προϊόντων. Υπάρχει το παράρτημα 4 με τα πολύ ευαίσθητα προϊόντα. Ούτω ή άλλω. Αυτό είναι ο βασικό λόγο που πιστεύουμε ότι ο κατάλογο πρέπει να παραμείνει στον τομέα των τεχνικών προδιαγραφών που αρχικά στοχευόταν ούτω ή άλλω. Ένα παράδειγμα. Και ο συναδελφό μου, ο κύριο Πούλμαν, το σχολίασε για την κρυπτογράφηση. Η κρυπτογράφηση των 48 bet και των 46 είναι των 64 μάλλον και 48 bit είναι κάτι που μπορεί να το μάθει και ένα 12χρονο σήμερα στο σχολείο. Ναι, εάν ο κατάλογος δεν είναι σωστός σε επίπεδο τεχνικών προδιαγραφών και δεν έχουμε το κατάλληλο επίπεδο τεχνολογίας, σε ένα χρόνο θα έχουμε ήδη πρόβλημα με τους ελέγχους. Γι' αυτό είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη και ο στόχος. Πάντοτε είναι διπλή και διτή η χρήση και ο σκοπός. Όλα αυτά μπορούν να, να χρησιμοποιηθούν στραβά και θα πρέπει να περιοριστούμε σε αυτού του είδους τα τεχνολογικά μέσα που πραγματικά μπορεί να είναι βλαβερά στην εποπτεία του κυβερνοχώρου το πρόβλημα είναι ότι ό,τι σε βλάπτει μπορεί να σε και καλύτερο. Αυτό είναι και η δυτή φύση του ίδιου του προβλήματος με τις ε, κυβερνοτεχνολογικές λύσεις. Μια απάντηση προς τον κύριο Φιέλνερ ίσως. Από όσα ξέρω και από αυτά που εγώ θεωρώ για το τι επιπτώσεις θα υπάρχουν στην κρυπτογράφηση έχουμε ξεκάθαρες αποδείξεις ότι ήταν επιζήμιο για την ευρωπαϊκή βιομηχανία για ένα διάστημα. Ξέρω ότι δεν μας αρέσουν πολύ οι αλλά κάναν κάτι πολύ σωστό με τον έλεγχο της ε, κρυπτογράφησης. Ξέρετε ότι σχεδόν όλη η τεχνολογία κρυπτογράφησης και τα ε, αντικείμενα κρυπτογράφησης μπορούν να πουληθούν σε όλο τον κόσμο, σε οποιαδήποτε χώρα είναι εξαιρέτω, με την εξαίρεση μόνο πέντε, τις οποίες δεν θέλω εδώ να ονομάσω και να κάτω ονομάσω. Γιατί ε, μήπως θέλουμε το ίδιο και εμείς ε, να κάνουμε με άλλε τεχνολογίες. Οι αμερικανικές εταιρείε, ακόμη και σήμερα, στην ε, ε, παρακολούθηση και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο είναι νούμερο ένα Θέλουμε να χάσουμε και άλλη καινοτομία και άλλες εταιρείες από την Ευρώπη προσπαθώντας να προστατεύσουμε τα θεμελιώδη δικαιώματά μας, διότι είναι σημαντικές αυτές οι τεχνολογίες και για αυτό το σκοπό. Και ένα βήμα προς την τελευταία ερώτηση που τέθηκε. Εάν θα θέλαμε λιγότερη καινοτομία και λιγότερο κέρδος. Επειδή η στρατηγική της εταιρείας μας είναι να κάνουμε και τους ανθρώπους να ζουν κάπως καλύτερα, να λιγοστέψει ο πόνος στον υπόλοιπο κόσμο. Οι τεχνολογικές λύσεις σκοπό έχουν και να προστατεύσουν τις ζωές των ανθρώπων, όχι απλώς τον ιδιωτικό τους βίο και τα δεδομένα τους. Αυτά τα δύο πάνε χέρι-χέρι. Άρα λιγότερη καινοτομία λόγω χάρη στον τομέα της υγείας είναι οπωσδήποτε όχι η απάντηση. Και βεβαίω θα πληγεί το κέρδο τη καινοτομία, αλλά δεν θα έπρεπε να είναι η επιλογή καινοτομία ή ανθρώπινα δικαιώματα. Θα έπρεπε να πηγαίνουν χέρι-χέρι. Και περισσότερη καινοτομία και περισσότερα ανθρώπινα δικαιώματα. Και λιγότεροι παραβάτε. Αυτή είναι η λογική μα και αυτό έχουμε έρθει εδώ να συζητήσουμε. Δεν πρόκειται να υπάρξει ούτε μία εταιρεία που θα έρθει εδώ να σας μιλήσει ή με την οποία μπορείτε να έρθετε σε επαφή στην καθημερινή σας ζωή που θα σας πει Α, θέλω πιο πολλά λεφτά, αλλά λιγότερα ανθρώπινα δικαιώματα. Ω ε, πολίτη που εργάζεται για εταιρεία, δεν το πιστεύω αυτό. Ευχαριστούμε ο κύριο Πούλμαν. Ευχαριστώ πολύ. Εκτιμώ τις ανησυχίες σας για το κατά πόσο μπορώ να βοηθηθώ και να κοιμάμαι καλύτερα τα βράδια και θα σας πω ότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η σαφήνεια. Το catch all να χρησιμοποιηθεί εκεί που η τεχνολογία προχωρά υπερβολικά ίσως γρήγορα. Η πολιτική δίνει την εντύπωση ότι δεν μπορούμε να νομοθετήσουν για κάτι που υπάρχει σήμερα και που μπορεί να μην υπάρχει αύριο. Δεν έχουμε δει ακόμα τις κατευθυντηρίες γραμμές. Το SDG διαδικασία υπάρχει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προτείναμε στην Επιτροπή να μιλήσει με τους φορείς τυποποίησης. Στον κόσμο της τεχνολογίας, των επικοινωνιών και της πληροφορικής υπάρχουν διάφοροι φορείς τυποποίησης, standardization, που καθορίζουν τεχνολογίες σε πολύ τακτά χρονικά διαστήματα και δεν έχουν ληφθεί καθόλου υπόψη. Και μετά τους έρχονται κατευθυντήριες γραμμές και είναι δύσκολο να ε, διατηρήσουμε την ε, εμπιστοσύνη μας για τη διαδικασία Κατσόλ, γιατί μας φαίνεται ως φενάκι, ως βιτρίνα για να καλύψει την ανεπάρκεια της προετοιμασίας των ε, νομοθετούντων. Είναι σημαντικό για μας να είμαστε μια γερμανική εταιρεία κυβερνοασφάλειας. Στο Άχεν έχουμε εξαιρετική πρόσβαση σε, στους ανθρώπινους πόρους, στο προσωπικό. Έχουμε νόμους που προστατεύουν πάρα πολύ την ιδιωτική σφαίρα και αυτό είναι επιχειρήματα πολύ σημαντικά. Είναι τεράστιο μάρκετινγκ τα τελευταία χρόνια για όλη τη βιομηχανία και κυρίως για την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Όταν ε, ισχύσει αυτός ο κανονισμός δεν σημαίνει ότι θα αλλάξω έδρα, αλλά θα πρέπει να ξοδέψω περισσότερους πόρους υποβάλλοντας συνέχειες αιτήσει για να κοιμάμαι καλύτερα το βράδυ και να πλημμυρίζω τον κύριο Πιτς και το γραφείο του με ερωτήσεις, ε, κάτι το οποίο θα αυξήσει τη γραφειοκρατία. Εμείς συζητούμε dual use filings για κρύπτο, για διαβατήρια, για θέματα μετανάστευσης. Μιλούμε για ψηφιακά διαβατήρια με κρυπτο το γράφηση εντός και αυτό θα μπορούσε να, να σημαίνει καταπίεση. Αυτό δεν ισχύει μόνο για τα ψηφιακά διαβατηρία. Αν θέλει κανείς και να καταπιέσει μπορεί να το κάνει και με τα αναλογικά διαβατηρία. Επομένως ζητώ από τη γερμανική κυβέρνηση να μου δώσει άδεια και θα δούμε με την Ομοσπονδιακή κυβέρνηση και τα τυπογραφία και τους εκδότες πώς θα γίνει. Ναι. Θα ήθελα εκεί να προσπαθήσω περισσότερο και λιγότερο με το να συμμορφούμε με όλα αυτά τα γραφειοκρατικά. Ε, και γι' αυτό έχω ενστάσεις για την πρότασή σας. Θα ήθελα επίσης να σας διορθώσω για κάτι. Η παράδοση της υπηρεσίας ε, ε, από την εταιρεία μου έγινε σε, σε, πελάτη εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος μετά την εξήγαγε και τη μεταπόλυσε αλλού. Η συμφωνία ποτέ δεν ολοκληρώθηκε, σταμάτησε 9 μήνες πριν επιβληθούν οποιασδήποτε κυρώσεις. Αυτή είναι η χαρακτηριστική βραδίτητα της πολιτικής διαδικασίας. Και τώρα μετακυλίουμε ακόμα πιο βαρύ καθεστώς της εταιρεία. Θα πρέπει οι εταιρείε από μόνες τους τώρα να αξιολογήσουν γρηγορότερα τους κινδύνους από μόνες τους. Εγώ είμαι υπέρ της εναρμόνισης Ευρωπαϊκή Ένωση της νομοθεσίας απολύτως. Αλλά ε, αν πρέπει να διαβάσω την κρυστάλλινη σφαίρα και να σας πω πόσο σίγουρο ένα συγκεκριμένο νομοθετικό καθεστώς θα αλλάξει την πολιτική των εταιριών για χή προϊόν ψηφιακό τεχνολογίας, ε, δεν μπορώ να το κάνω. Ευχαριστώ πολύ. Στρέφουμε τώρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να υποβάλει τα τελικά σχόλια για τη συζήτηση αυτή. Ο αρμόδιος διευθυντής ε, υπεύθυνος για το εγχείρημα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είναι αδύνατο σε πέντε λεπτά να αντιδράσουμε σε όλα αυτά τα ζητήματα που έχουν τεθεί σήμερα το απόγευμα από ε, τους εμπειρογνώμονες και τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το καλύτερο που θα έπρεπε να κάνω και θα προσπαθήσω να κάνω είναι να αναφερθώ σε ορισμένα ζητήματα και να πω δύο λόγια για τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει το ζήτημα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ποια είναι η νοοτροπία που τη χαρακτηρίζει, ποιο είναι ο συλλογισμός πίσω από την πρόταση του Σώματος των Επιτρόπων προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα συνεχίσουμε να ενημερώνουμε τους συνομοθέτες για να προχωρήσει η νομοπαρασκευαστική διαδικασία. Να εστιάσω την προσοχή μου σε δύο-τρία ζητήματα λοιπόν. Πρώτον, για το θέμα της εισαγωγής της διάστασης της ασφάλειας που είναι μια αυτόνομη διάσταση. Είναι ένα θέμα πολιτικού κατοφλίου, threshold είναι αυτό που αποφάσισε να διαγράψει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρότασή της. Είναι μια σταθμισμένη ε, διάσταση και θα υπάρξουν συζητήσεις για το βελινεκές. Άκουσα αυτά που είπε από την Βάφα για τη διατύπωση των κριτηρίων στο, ε, ε, κάτω από το 1β και 1α. Όμως είναι μια διάσταση και νομίζω ότι υπόθηκε από τους ομιλητές που θα συμβάλλει στο να εξισώσουμε τους όρους του παιχνιδιού για όλες τις επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια και αυτό είναι πολύ σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως θεσμικό όργανο και πρέπει να είναι και πρέπει να σχεδιαστεί με τρόπο αναγκαστικά που δεν επιτρέπει παραθυράκια και κενά σε ένα περιβάλλον όπως το ψηφιακό που αλλάζει τόσο γρήγορα. Και γι' αυτό αυτό θα διαμορφώσει και το πιο βεληνικές θα έχει η πρόταση φιλόδοξο ή όχι. Ε, πολλοί στη συζήτηση εστίασαν την προσοχή τους στην ανάγκη για μεγαλύτερη σαφήνεια, μεγαλύτερη ακρίβεια στην νομοθετική πρόταση. Αυτός είναι και ο σκοπός των κριτηρίων που προτείνουμε θα υπάρξει κατά πάσα πιθανότητα ανάγκη να αναπτύξουμε και να μελετήσουμε περισσότερο την εφαρμογή των κριτηρίων, ταυτοποίηση των δημοσίων φορέων, πρακτικές λεπτομέρειες εφαρμογής για τον εντοπισμό σοβαρών παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καταστάσεις συγκρούσεων, ε, κυρώσεις, κατασταλτική διαδικασία. Όλα αυτά πρέπει να τα αναπτύξουμε έτσι περαιτέρω. Από δική μας πλευράς ξέρετε ότι πιστεύουμε ότι αυτή η δουλειά εμβάθυνσης που είναι επιχειρησιακή, λειτουργική, εκφύσεως, άρα πρέπει να είναι αρκετά ευέλικτη, ούτω ώστε να μπορεί να είναι αποτελεσματική, μπορεί να πάρει τη μορφή των κατευθυντήριων γραμμών με επιτυχία. Και αντιδρώ και απαντώ στον κύριο Πούλμαν λέγοντας ότι η ακρίβεια και η σαφήνεια θα έρθει μόλις δεσμευτούν τα θεσμικά όργανα, δηλαδή αναλάβουν τη τεχνική δουλειά για να υπάρξουν κατευθυντηρίες γραμμές και έτσι το συμβόλαιο να μπορούμε να το έχουμε ολόκληρο και όχι μόνο τις μισές του σελίδες. Ας δεσμευθούν οι συνομοθέτες να δουλέψουν πάνω σε αυτό για να καθαρίσουμε με ακρίβεια τις κατευθυντήρες γραμμές σε τεχνικό επίπεδο. Τώρα, καθήκοντα των επιχειρήσεων θα είναι να διεξάγουν δράσεις για τη φυσιολογική, κανονική, δέουσα επιμέλεια, όπως προβλέπεται από την υφιστάμενη νομοθεσία. Δεν είναι κάτι το ασυνήθιστο και ακριβώς ε, λόγω αυτού δεν μας πείθουν οι ανησυχίες που εκφράστηκαν στη συζήτηση ότι η έλεγχη για την ανθρώπινη ασφάλεια θα οδηγήσουν σε ένα κατακλυσμό αιτήσεων αδειοδότησης. Δεν πιστεύουμε εμείς ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο. Και τρίτον, για το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την κυβερνοασφάλεια, να πω και δύο λόγια για τη διαπίστωση σύμφωνα με την οποία η ανάπτυξη των ελέγχων σε αυτό το τομέα αντιβαίνει και αντίκειται στη συμφωνία ITA. Από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής εμείς πιστεύουμε ότι το γεγονός ότι μια τέτοια συμφωνία θα εξαλείψει δασμού σε, μεγάλα, σε πάρα πολλά προϊόντα δεν μπορεί να μπει σε μια ζεγαριά και να ισοσταθμιστεί με την ανάγκη να ελεγχθούν ε, ορισμένα πολύ μικρότερα σε όγκο και σε μέγεθος και σε αριθμό προϊόντα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια. Είναι απαραίτητο να συνεχίσουν να συνυπάρχουν τα δύο. Ένα δεύτερο ζήτημα που είναι χρήσιμο να θίξει κανείς είναι οι ανησυχίες για τη διευκρίνηση των ελέγχων σε σχέση με την τρομοκρατία. Και επιμένω στον όρο clarification, διευκρίνηση, διασάφηση, γιατί είναι ε, ε, πολιτική που εφαρμόζεται από τα κράτη-μέλη και όχι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα μέλη στο Βάσεναρ υπογραμμίζουν τη σημασία όλων αυτών. Άρα υπάρχει προσανατολισμός πολιτικός, ε, υπάρχουν γενικές κατευθύνσεις, πολιτικές γραμμές για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και είναι δύσκολο από τη μία να λέμε ότι είναι πολιτική προτεραιότητα η τρομοκρατία και από την άλλη να έχουμε κανονισμό, να συνεχίσουμε να έχουμε κανονισμό που δεν λαμβάνει υπόψη του τα θέματα της τρομοκρατίας. Τώρα για το τράνζιτ, τη διαμεστακόμιση, την διαμεσολάβηση για τεχνική βοήθεια. Θα είμαι εξαιρετικά σύντομος και θα πω ότι από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν πιστεύουμε σε ένα σύστημα à la carte σε αυτή την περίπτωση, όπου κάθε κράτος μέλος θα αποφασίζει μόνο του κατά πόσο θέλει ή μπορεί να ελέγξει χύψη ή μορφές συναλλαγών. Εάν μια συναλλαγή δημιουργεί κίνδυνο, τότε πρέπει να ελέγχεται από όλα τα κρατημέλη. Αυτή είναι η άποψή μας και πρέπει να έχουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση κοινή προσέγγιση και κοινό μοίρα πλάσμα της ευθύνης για τους κινδύνους. Γιατί, και δεν πιστεύουμε ότι θα έχουμε ένα σωρό εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις διαμετακόμισης. Τέταρτον, για το ζήτημα της βελτιστοποίησης των πρωταπαιτούμενων για την αδειοδότηση, optimization, να πω, απαντώντας σε κάτι που είπατε και εσείς κύριε Πρόεδρε, απαντώ λέγοντας ότι είναι σημαντικό και καταλαβαίνουμε ότι για την κοινή προσέγγιση για την αδειοδότηση πρέπει να έχουμε building blocks και πρέπει για να τα έχουμε να καταλάβουμε το πώς λειτουργούν οι έλεγχες εξαγωγές και για να καταλάβουμε πώς λειτουργούν οι ε, έλεγχες εξαγωγές καλύτερα πρέπει να βελτιώσουμε το σύστημα πληροφόρησης που έχουμε και συλλογή στοιχείων. Άρα ολοκληρώνω με ένα τελευταίο σχόλιο που εκφράζω την έκπληξή μου που δεν αναφέρθηκε τον έλεγχο των ενδοευρωπαϊκών εμβασμάτων μεταφορών transfers, intra-EU transfers. Έχει τεθεί στο Συμβούλιο στον άλλο συνομοθέτη με την επιφύλαξη των ευαισθητησιών δύσκολα δικαιολογούμε ότι ο κατάλογος των ζητημάτων αυτών δεν έχει ενημερωθεί, δεν έχει επικαιροποιηθεί. Δύσκολα δικαιολογείται το ότι τα κράτη-μέλη ατομικά συνεχίζουν να δίνουν άδεια για κάθε διαφορετική συναλλαγή εξεχωριστά ατομικά εντός της ενιαίας αγοράς. Είναι δύσκολο αυτό να σταθεί δηλαδή. Πιστεύουμε κύριε Πρόεδρε ότι η πρόταση είναι ισορροπημένη. Σας ευχαριστούμε που, δώσαμε την, που μας δώσατε την ευκαιρία να συμβάλλουμε στη συζήτηση. Ευχαριστώ. Κύριε Μπούχνερ, θέλετε να κάνετε κάποιες τελευταίες παρατηρήσεις. Λίγες παρατηρήσεις. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ομιλητές, τους ειδικού και κυρίως την Κομισιόν για τον χρόνο τους. Η εντύπωσή μου είναι πραγματικά ότι είναι σαφές ότι απαιτείται μια μεταρρύθμιση αυτού του κανονισμού που αφενός θα ανταποκρίνεται στις νέες προκλήσεις της ε, ψηφιακής εποχής αλλά ταυτόχρονα θα έχει σαφείς ε, και εφαρμόσιμους ε, κανόνες για τις επιχειρήσεις στην Ένωση για να έχουν μια ασφάλεια προγραμματισμού. Και βεβαίως ε, συμφωνώ εδώ πέρα με τους εκπροσώπους του κλάδου. Τέλος, ε, θα ήθελα να πω πως ε, έχουμε ένα πολύ αυστηρό χρονοδιάγραμμα και νομίζω ότι θα μπορέσουμε να τα καταφέρουμε και εν πάση περιπτώσει η πόρτα μου είναι ανοιχτή για όλους τους συναδέλφους και τους ειδικού σας. Ευχαριστώ, ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους ειδικού μας. Ήταν πάρα πολύ επικοδομητική η επίσκεψή σας και μην διστάσετε να έρθετε σε επαφή ξανά μαζί μας ανα πάσα στιγμή. Ευχαριστώ πάρα πολύ.